Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Το σημείο 13 είναι ανταλλαγή απόψεων με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας και Εμπορίου του Κοινοβουλίου της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τις εκατέρωθεν εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις. Καταρχήν να, να παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας, ο κ. Τζον Χέις, εξ αριστερών μου, δεν θα πω πότε γεννηθήκατε. Θα διαβάσω τα στοιχεία που έχω για σας χωρίς την ημερομηνία γέννησή σας. Μισό λεπτό να το βρω μόνο. Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας και Εμπορίου. Στη συνέχεια ο Φιλ Γκόβ, τον Φιλ τον γνώριζα όταν ασχολούμεθα με διάφορες εμπορικέ συναντήσεις με τη Νέα Ζηλανδία, διότι τότε ήταν υπουργό Εμπορίου. Και ο Πολ Χάτσινσον που είναι στο ακροατήριο ήταν μαζί μας. Και είναι μαζί μας και ο Σούα Βίλιαμς. Τέσσερις προσκεκλημένους έχουμε. Επίσης, χαιρετίζουμε και τον πρέσβη Κύριε Βιτάλη. ο στόχο τη ε, συνάντησή μα είναι να συζητήσουμε τι εμπορικέ και επενδυτικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Νέα Ζηλανδία, ε, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα και να εξετάσουμε την εταιρική μα σχέση από μια ευρύτερη περιφερειακή άποψη. Και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι ο ανοιχτό χαρακτήρα τη Νέα Ζηλανδία στο διεθνέ εμπόριο ε, καλύπτει διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων και διάφορες συμφωνίες FTA με την Κίνα, την Ινδία, την Ταϊβάν, Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν υπό διαπραγμάτευση. Τελωνιακή Ένωση, η Νέα Ζηλανδία εξετάζει εταιρικές σχέσεις και ολοκληρωμένες εμπορικές σχέσεις με την Ασία. Φαντάζομαι ότι το TPP θα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή. Έχουμε πολλά να διδαχθούμε στην Ευρώπη από τις εμπορικές σας πολιτικές, όπως επίσης και από τις συμφωνίες σας για το εξωτερικό εμπόριο της FTA που προαναφέραμε. και για την γεωργία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ε, όπως και για την μεταρρύθμιση της γεωργίας και υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας μέσω διαπραγματεύσεων, συμφωνία πλαίσιο ε, ξεκίνησε το καλοκαίρι και ελπίζουμε ότι ε, θα υπάρξουν πολλά εμπορικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου ενέκρινε την τροποποιητική διμερή συμφωνία για την ε, έγκριση τύπου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας. Θέλω να σας δώσω το λόγο κατευθείαν γιατί ε, οι συνάδελφοι θέλουν να ακούσουν αυτά που εσείς έχετε να πείτε. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο, ιδιαίτερα στην οικονομική θέση που βρισκόμαστε. Και πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι πάντοτε καλύτερη λύση από την βοήθεια. Και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στο εμπόριο. Εσείς, ιδίως με την κοινή γεωργική σας πολιτική πριν από ορισμένα χρόνια, εν μια νυχτή δημιουργήσατε τεράστια πρόοδο. Ο κύριος Εξαριστερών, ο κύριος Γκόφ ε, ήταν ε, αυτός ε, που το ε, επιτέλεσε. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για το μέλλον. Μικρόφωνο παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε για να μπορέσουμε ε, να εκφράσουμε τις απόψεις της αντιπροσωπείας μας εδώ στην Ευρώπη. σε μια συνεδρίαση της ΑΣΕΜ τον περασμένο μήνα εκφράσαμε αυτές τις απόψεις μαζί με την Αυστραλία και τη Ρωσία ήμασταν παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση ΑΣΕΜ εξετάσαμε διάφορα θέματα ε, και έβλεπα τους Ευρωπαίους εταίρους στη συνεδρίαση και σκεφτόμουν ότι ίσως οι Ευρωπαίοι να νομίζουν ότι εμείς ε, γυρίζουμε την πλάτη μας ε, στην Ευρώπη και θέλω να τονίσω ότι εμείς κατά κανένα τρόπο δεν στρέφουμε την πλάτη μας στην Ευρώπη και μάλιστα θα είμαι υπεύθυνο μιας διακομματικής αντιπροσωπείας από τη Νέα Ζηλανδία στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα και πραγματικά υλοποιούμε σήμερα εκείνη την ε, ε, υπόσχεση που δώσαμε σε εκείνη τη συνεδρία πριν από ένα μήνα. Χαιρετίζουμε την ευκαιρία σε επίπεδο βουλευτών να έρθουμε σε στενότερη επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωριστά. Σήμερα το πρωί ήρθαμε από τη Δανία και θα επισκεφθούμε και άλλες δύο πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Στο παρελθόν και άλλοι συνάδελφοι έκαναν καλές ε, επικοδομητικές συναντήσεις και νομίζω ότι σήμερα έχουμε μια καλή ευκαιρία να συναντηθούμε σε επίπεδο Επιτροπής Εμπορίου εδώ στις Βρυξέλλες. Και ελπίζω ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι η πρώτη συνάντηση που θα ξεκινήσει μια σειρά άλλων παρόμοιων συναντήσεων απέχουμε 27 ώρες πτήσης ε, η Ευρώπη από τη Νέα Ζηλανδία. Παρ' αυτά η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι δύο πολιτισμοί που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά έχουμε πολύ παρόμοιες αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το περιβάλλον, για το εμπόριο. Ξέρουμε ότι μπορούμε να συνομιλούμε απευθείας γιατί έχουμε αυτές τις κοινέ αξίες. Και πιστεύουμε ότι η επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδου σημασίας. Θυμάμαι όταν ως διπλωμάτης συνόδευα Υπουργού, σε επισκέψεις τους ε, όταν έρχονταν για προσκύνημα εδώ στην Ευρώπη. Θυμάμαι ε, ότι όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας έγιναν ακόμη σημαντικότερα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική εμπορίου. και ιδιαίτερα ε, μετά τον Ιούλιο και την καταψήφιση της Συμφωνίας Άκτα, νομίζω ότι αυτό άλλη μια φορά καταδεικνύεται. Φαίνεται η σημασία την οποία έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας συγκεκριμένα όσον αφορά τη θέσπιση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμεί ω βουλευτέ που μιλούν σε βουλευτέ κατανοούμε την σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το εκτιμούμε ιδιαίτερω. Είμαστε μια μικρή χώρα που εξαρτώμεθα από το εμπόριο. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Νέα Ζηλανδία και αυτό πάντοτε ίσχυε και θα συνεχίσει να ισχύει, είμαι βέβαιος. Καταρχήν, διότι είναι σημαντική αγορά. Για μας είσαστε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά μετά την Αυστραλία, την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες ιστορικά ήταν η πιο σημαντική αγορά για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά έχει μειωθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λόγω της αύξησης της σημασίας ε, της Ασίας και λόγω της διαφοροποίησης. Το θέμα της διαφοροποίησης νομίζω ότι το γνωρίζετε στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ο κύριος Γκόφ εδώ εξ αριστερών μου ήταν ε, υπεύθυνος της εμπορικής πολιτικής, ήταν σε μια κυβέρνηση ε, που ε, είχε αναλάβει μια κατάσταση οικονομικής κρίσης. Και εν μια νυχτή μεταρρυθμίσαμε τη γεωργία και όλες τις γεωργικές επιδοτήσεις, γιατί δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή παρά να το κάνουμε και αναγκάστηκαν οι παραγωγοί μας να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και τις αγορές τους και ως ερετός βουλευτής σε ένα κοινοβούλιο από αγροτική εκλογική περιφέρεια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η έκθεσή μας στη διεθνή αγορά ε, αύξησε πάρα πολύ την παραγωγικότητα στον τομέα της γεωργίας. Πολύ περισσότερο από ότι τα ωφέλη τα οποία είδαμε στον τομέα της μεταποίησης. Η γεωργία παραμένει βασικό τμήμα του εμπορικού μας χαρτοφυλακίου. Όταν μιλάμε όμως για την γεωργία στη Νέα Ζηλανδία σήμερα, μιλάμε για πολύ ευρύτερες υπηρεσίες και αγορές από ό,τι στο παρελθόν. Και πολλές από αυτές τις νέες αγορές βρίσκονται στην Ασία λόγω της εγκύτητός μας προς την Ασία και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της περιφέρειας της Ασίας. Θα συνεχίσουμε την εξάπλωσή μας στην Ασία με συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Ο Φιλ Γκόφ ε, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία εμπορική με την Κίνα και είμαστε και η πρώτη χώρα του ΩΣΑ που έκανε μια τέτοια συμφωνία. συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και με την ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο ε, της ε, οικονομικής συνεργασίας ε, του ειρηνικού και ως μεγαλύτερη οικονομική ενότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Έχει, κλείσει, έχει συνάψει μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κορέα και έχει και διαπραγματεύσεις με άλλες ασιατικές χώρες. Συζητώντας όμως ε, τα ωφέλη, το, να συζητάμε τα ωφέλη μιας τέτοιας πολιτικής δεν είναι το βασικό θέμα. Το βασικό θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για το εμπόριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία έχουν κάποια κοινά γνωρίσματα. Το βασικό κοινό γνώρισμα είναι η κοινή μας δέσμευση υπέρ ανοιχτών κανόνων και δίκαιων κανόνων και έχουμε επωφεληθεί από τους δίκαιους αυτούς κανόνες και η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Ζηλανδία όπως και πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών της ΓΑΤ και πολύ συχνά ηγούμεθα διαπραγματεύσεων στο διεθνές εμπόριο. για πολλούς οι καθυστερήσεις και η στασιμότητα του γύρου της Ντόχα είναι απογοητευτικές και μάλιστα εμείς θεωρούμε ότι είναι και ανησυχητικές. Συγκρίνοντας λοιπόν τον αριθμό των ε, εμπορικών συμφωνιών δεν καταλήγουμε πουθενά. Χρειαζόμαστε κοινού κανόνες, διαφορετικά τα ωφέλη από αυτές τις FTAs, από αυτές τις εμπορικές συμφωνίες δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας βασικός φορέας για το διεθνές εμπόριο όσον αφορά αυτούς τους κανόνες και μπορεί να διαφωνούμε σε ορισμένα θέματα. Σε γενικές γραμμές όμως πάντοτε επωφελούμεθα από την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πολυμορφία και από τα κοινά μας χαρακτηριστικά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νοιάζεται όσο και εμείς για την πρόοδο του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ικανότητα να ηγείται και θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγείται. Στην Ασία χρειαζόμαστε την ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τις δικές της συζητήσεις με τις μεμονωμένες χώρες και αυτό το χαιρετίζουμε παρότι μπορεί να μην είμαστε εμείς μία από τις χώρες αυτές. Ελπίζουμε ότι μεσοπρόθεσμα θα συμμετάσχουμε και εμείς αλλά οι διμερείς συζητήσεις ε, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις συνολικές ε, ε, συζητήσεις που θα οδηγήσουν στο να τηρούνται ορισμένοι κανόνες από τις συμβαλόμενες χώρες. Εδώ ακριβώς έχουν ένα κοινό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία στο εφαρμόζονται δηλαδή αυτοί οι δημοκρατικοί κανόνες από όλες τις χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τις κοινοβουλευτικές μας παραδόσεις. Εμείς χαιρετίζουμε τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επαφές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιφέρειά μας και θα θέλαμε να εξερευνήσουμε και άλλους τρόπους κατά τους οποίους θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να το επιτύχουμε. Ας υποστηρίξουμε η μεν δε για να ενθαρρύνουμε και να διδάσκουμε οι μεν δε και να βελτιώνουμε την περιφερειακή μας οικονομική συνεργασία ώστε να οδηγηθούμε στην της πολυμερής σχέσεις μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά και αν ε, κρατήσετε μία σκέψη από όλα αυτά τα οποία σας είπα, θα ήθελα να σας πω ότι στην άλλη άκρη του κόσμου η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία είναι φίλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Ειρηνικό. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι σχέσεις μεταξύ των κοινοβουλίων μας. Είτε συναντιόμαστε εδώ στις Βρυξέλλες, είτε συναντιόμαστε κάπου στην Ασία, είτε στη Νέα Ζηλανδία. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι επαφέ. Σα ευχαριστώ πολύ και εκ μέρου τη αντιπροσωπεία μας σα ευχαριστώ πολύ που μα καλέσατε και αν έχετε ερωτήσει, ευχαρίστω θα σα απαντήσουμε. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζον. Ήδη έχω κατάλογο μελητών, αλλά δεν ε, ξέρω αν κάποιος άλλος από την αντιπροσωπεία που έχει έρθει εδώ θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να γνωρίζετε ότι η Νέα Ζηλανδία είναι πάρα πολύ μακριά. 18.000 χιλιόμετρα είμαστε μακριά από την Ευρώπη. Όμως ε, πολλές από... Συχνά η προέλευσή μας σε μεγάλο βαθμό είναι από την ε, Ευρώπη και για τις αξίες μας το λέω αυτό και ήμασταν πάντοτε σε σχέση συνεργασίας ε, όταν ήρθα σε επαφή με την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε διαφορές παρά τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση. Έχουμε μεγάλη δυσκολία να διαφωνήσουμε με τους στόχους και τις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είμαστε εδώ για την επέτειο της ε, εκεχηρίας ε, για μία περίοδο ε, χάθηκαν 180.000 Νεοζηλανθοί μιλάμε για μία χώρα ε, που έχει πληθυσμό κάτω του 1 εκατομμυρίου είμαστε οι, σας, οι μεγαλύτεροι σας υποστηρικτές στην, σε μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπάρχει πια πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το λέω αυτό από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί εμείς ε, είχαμε συμπατριώτες που έχασαν τη ζωή τους, αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους ε, για το ευρωπαϊκό έδαφος. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσω λέγοντας ορισμένα πράγματα που είπε και ο συνάδελφος. Ε, είμαστε υπέρμαχοι του πολυεθνισμού, ήμουν στη Γενέβη πριν από τέσσερις, τέσσερα χρόνια, στο πράσινο δωμάτιο, σε διάσκεψη του ΠΟΕ, που φτάσαμε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε ε, το γύρο της Δόχα. Ήταν μια τραγωδία για όλες ε, τις χώρες του κόσμου, αλλά ειδικότερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την συμφωνία αυτή και θα ήθελα να επενέσω την ε, σχέση συνεργασίας ε, που είχαμε τον Πίτερ Μάντελσον τότε που ήταν ε, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να κινηθούμε προς την άρση των εμποδίων των εμπορικών μεταξύ των χωρών όχι μόνο μέσω διμερών εμπορικών συμφωνιών αλλά και με έναν τρόπο που μπορεί μόνο παγκόσμια Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου να κάνει. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Βέβαια μπορεί να μας πάρει πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε περάσει εντωμεταξύ σε ζώνες ελευθέρου εμπορίου, σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Ε, και μάλιστα ο Βαγγέλης Βιτάλης, ένας από τους συναδέλφους μου που, ε, τους συναδέλφους μου που είναι ο πρέσβης της Βρυξέλλες, ε, είναι υπεύθυνο διαπραγμάτευσης, μια περιεκτική συνεργασία μεταξύ της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των χωρών ΑΣΕΑΝ. Είναι μια υψηλού επίπεδου ποιότητα, η, συγγνώμη, συμφωνία, η οποία συμπεριλαμβάνει εμπορικές και ε, πτυχές συνθήκων εργασίας και περιβαλλοντικές πτυχές ε, και πρόκειται για μια συμφωνία η οποία ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Μία ακόμη που, ε, συμφωνία που υπογράψαμε τον Απρίλιο του 2008, μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα. Είμαστε η μόνη χώρα ε, ΑΣΕΑΝ ε, που έχει τέτοιου είδους συμφωνία αφορά το 98% των δασμών, ε, καλύπτονται το ε, τομείς όπως το εμπόριο, ε, η εργασία και το περιβάλλον. Τέσσερα χρόνια μετά έχει τριπλασιαστεί, έχουν, έχουν τριπλασιαστεί εξαγωγές μας στο, στη, με την Αυστραλία, με τη, σύνο, με την Κίνα, οπότε σε όλες αυτές τις συμφωνίες ε, ε, που, με τις οποίες συμμετείχε η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, ε, και η Χιλή διευρύνθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν τον Μεξικό και άλλες χώρες. Ε, στην Ασία ε, υπήρχε λοιπόν ε, μία πληθώρα συμφωνιών εμπορίου, όμως υπήρχε και κάποια στρέβλωση στην περιφέρεια λόγω όλων αυτών των συμφωνιών και ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα συμμετέχει περισσότερο στο εμπόριο με την Ασία και εμείς ως φιλικά προσκύμενοι προς την Ευρώπη χώρα μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, και να έχουμε ε, διαπραγματεύσεις ε, με τις χώρες ΑΣΕΑΝ την Αυστραλία ε, δηλαδή τη Νέα Ζηλανδία, τις χώρες ΑΣΕΑΝ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Είναι σημαντικό να υπάρχει ε, με την περιφερειακή εμπορική συνεργασία που θα συμπεριλάβει την Ινδία, ε, την Κίνα, την Κορέα και την Ιαπωνία, είναι σημαντικό να μην ε, υπάρχει διάκριση εναντίον, τας, σας ε, όταν προσπαθείτε να γίνετε η μεγαλύτερη και πιο ραγδαία αυξανόμενη οικονομία στον κόσμο. Όταν κάποτε ήρθαν οι Υπουργοί Νεοζηλανδοί στην Ευρώπη για να αγωνιστούν για τις εμπορικές συμφωνίες που είχαμε με το Βασίλειο, γιατί εγώ όταν ήμουν παιδί οι περισσότερε εξαγωγέ μας πήγαιναν εκεί. Ήταν μια τραυματική εμπειρία για τη Νέα Ζηλανδία. Να σας πω την αλήθεια, πιστέψτε με, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, ήταν πάρα πολύ ε, τραυματική εμπειρία. Και τη δεκαετία του 80, όταν πρώτη φορά ανέλαβα καθήκοντα υπουργού, αλλάξαμε τη χώρα μας ε, από μια χώρα που έμοιαζε πολύ με τις πρώην ε, ανατολικές οικονομίες, ε, τις μετατρέψαμε σε μια από τις πιο ελεύθερες και ανοιχτές οικονομίες του κόσμου. Δεν υπήρχαν επιδοτήσεις πλέον σχεδόν μια νυχτή τις καταργήσαμε. Το σύστημα, για την γεωργία μιλάω, γιατί οι επιδοτήσεις κατέστρεψαν την γεωργία, γιατί η γεωργία ε, παρήγαγαν για την επιδότηση και όχι για τα προϊόντα. Άλλαξαν αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Οι γεωργοί μας τώρα συναλλάσσονται με τον κόσμο χωρίς καμία απολύτως επιδότηση. Δεν υπάρχουν επιδοτήσεις που να στρεβλώνουν οτιδήποτε την παραγωγή τους ε, και ε, τελικά ε, παράγουν ε, ε, γεωργικά προϊόντα με τη γη τους και μάλιστα με περιβαλλοντικό τρόπο, με ιδιαίτερα περιβαλλοντικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε και να βαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τις εμπορικές μας σχέσεις, μια και πρόκειται για χώρες που έχουν τόσα πολλά κοινά. Κάποτε, και αυτό είναι το τελευταίο που θα πω, η Ευρώπη φοβόταν τη Νέα Ζηλανδία και τη γεωργική της παραγωγή. Ε, τώρα είναι τόσο διαφοροποιημένη η παραγωγή μας που δεν είμαστε καμία απειλή για τους γεωργούς στην Ευρώπη. Θέλουμε σε ισότιμη βάση να συναλλαζόμαστε, όπως όλα τα προϊόντα σας έρχονται στη Νέα Ζηλανδία χωρίς ε, δασμούς ε, πάνω κάτω. Θα θέλαμε το ίδιο να ισχύει, το ίδιο και για τα δικά μας προϊόντα όταν αυτά εισέρχονται στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Φιλ. Έχεις απόλυτα δίκιο. Ήμουν και εγώ στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τότε που ασχολούμεθα με τα θέματα των αγροτών και διευκολύναμε το πεδίο στις διαπραγματεύσεις τότε. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον Πολ Χάτσινσον, ε, μέλος της ε, Επιτροπής Εμπορίου και ε, Άμυνας και Υγείας. θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι θα αρχίσουμε την ψηφοφορία στις 4. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Χάτσινσον. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερω ε, την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι εδώ στην Ευρώπη. Και εγώ είμαι από μια αγροτική εκλογική περιφέρεια, όπω και ο συνάδελφο, και ένα από τα χαρακτηριστικά τη περιφέρειά μα είναι ότι είμαστε η μεγαλύτερη παραγωγή κρεμμυδιών στη Μεγάλη Βρετανία και το 50% αυτών των κρεμμυδιών εξάγονται στην Ευρώπη. Όπως και οι συναδελφοί μου λοιπόν, θέλω να πω ότι μία είσοδος σε μια τέτοια αγορά που έχει τεράστια σημασία για μας, όπου ε, δεν έχουμε δασμούς, θα θέλαμε να έχουμε κάποιους δασμούς για τους αγρότες μας, ε, και για τους αγρότες μας είναι πολύ πιο δύσκολο το να έχουν να ξεπεράσουν άλλο ένα φραγμό όπως είναι οι δασμοί. Υπάρχουν και πολιτιστικοί και οικονομικοί δεσμοί με την Ευρώπη. Αλλά και πιο πρόσφατα έρχονται στην Ευρώπη πολλοί Νεοζηλανδοί για κάποια χρόνια, όπως ήρθα και εγώ μετά τις σπουδέ μου, για μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασία και μετά επανέρχονται στη Νέα Ζηλανδία. Υπάρχει μία έντονη ανταλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών και εργαζομένων με τη Νέα Ζηλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις σχέσεις μας γιατί ακριβώς αυτές ε, οι πολιτιστικές και ιστορικές αξίες αποτελούν τη βάση συνεργασίας των χωρών μας. Προσπαθούμε να έχουμε διαφοροποιημένο παγκόσμιο εμπόριο και αυτές τις πολιτιστικές και ιστορικές αξίες. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι στη Νέα Ζηλανδία εκτιμούμε ιδιαίτερα το όραμα της ευρωπαϊκής κοινότητας το όραμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη, για τις αξίες, για όλους. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε εμείς από μακριά, στην άλλη άκρη του κόσμου, στο νότιο ειρηνικό. Και όταν βλέπουμε ότι λειτουργεί το δικό σας σύστημα, είναι κάτι το οποίο θα θέλουμε να εφαρμόσουμε και εμείς και θα μπορούμε να το προτείνουμε ως πρότυπο σε άλλες χώρες στην Ασία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί όσο καλά θα θέλαμε. Και όπως είπε ο Φιλ υπάρχει μια πληθώρα συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, είμαι κάπως σε δύσκολη θέση όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποιες από τις χώρες εταίρους με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει εδώ μεγάλη δύναμη γιατί μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα μοντέλο κουλτούρας και δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την ευκαιρία που μας δίνετε να είμαστε σήμερα εδώ και προσβλέπουμε στις συζητήσεις που θα κάνουμε let me just uh, firstly greet and... Ο κύριο Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα εδώ και θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία λένε οι συναδελφοί μου, δηλαδή ότι την Ευρώπη ε, τη βλέπουμε με θαυμασμό και με έκπληξη, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικές προκλήσεις, πολύ περισσότερες από ό,τι άλλες χώρες. Το εμπόριο είναι σημαντικό κομμάτι ε, των λόγων για τους οποίους βρισκόμαστε εδώ, αλλά όχι ο μοναδικός. Εμείς που είμαστε φίλοι από την άλλη άκρη του κόσμου έχουμε και κοινές αξίες κοινέ αξίε στον τομέα του περιβάλλοντο και ο Ειρηνικό είναι μια περιοχή με την οποία έχουμε πολλέ σχέσει και ε, υπάρχουν πολλά ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και πολλά άλλα κράτη. Επίση μα απασχολούν θέματα περιφερειακή ασφάλεια. θα θέλαμε πολλές ε, μικρές ε, χώρες έθνη να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάποιους, κάποια προβλήματα σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Θεωρώ ότι ε, ήταν αυτό μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. Όπως ε, μπορούμε να υποφεληθούμε και εμείς από εσά, σίγουρα θα υπάρχουν αντίστοιχα ευκαιρίες από τις οποίες μπορείτε και εσείς να υποφεληθείτε. Ευχαριστώ πολύ και θα δω. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην Κότλιβ Χρυστριβιού, η οποία είναι υπεύθυνη των, ε, της ε, ε, Επιτροπής ε, για τις σχέσεις με την Νέα Ζηλανδία. Κυρία Κβίστου Τουροβόλη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί στο κοινοβούλιο μας ε, υπάρχει πολυγλωσία και θα μιλήσω γερμανικά. Χαίρομαι ε, και εγώ που είστε σήμερα κοντά μας. Και μάλιστα διότι όπως είπατε κι εσείς έχουμε κοινέ αξίες. Ε, είναι προφανές και δεν χρειάζεται καν να το επαναλάβω. ως υπεύθυνη της ε, ομάδας παρακολούθησης γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, προβλήματα. Θέλουμε να οικοδομήσουμε ακόμη καλύτερες σχέσεις και να αντιμετωπίσουμε όλες τις ε, δυσκολίες. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις καλές σχέσεις που ήδη υπάρχουν και σε αυτά που είπατε άκουσα κάτι πολύ σημαντικό για την ανταλλαγή νέων ε, μεταπτυχιακών σπουδαστών ή εργαζομένων. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα, πολύ συγκεκριμένα, μπορούμε να παράσουμε μεγαλύτερη υποστήριξη. Πολλοί ε, νεαροί Γερμανοί αυτή τη στιγμή θεωρούν τη Νέα Ζηλανδία ονειρεμένο τόπο διακοπών. Γιατί με το σακίδιο στην πλάτη φεύγουν γιατί στην αρχή φεύγανε για Αφρική, μετά Αυστραλία, τώρα της μόδας είναι η Νέα Ζηλανδία. Είσαστε στη Γερμανία η χώρα της μόδας. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω αυτό μπορώ να το πω εξ όλων των συναδέλφων, έχουμε και εμείς την ίδια πολυμερή προσέγγιση για το εμπόριο και για τις εμπορικές συμφωνίες. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε με, με τα λύπης ότι ο γύρος της Ντόχα δεν ε, έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό αυτή τη στιγμή και πολύ ρεαλιστικά μπορούμε να το δούμε σαν ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των διμερών και των πολυμερών συμφωνιών. Ακόμη και το ενδιάμεσο στάδιο δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί θετικό. Και θα επιθυμούσαμε να επιληθούν καλύτερα τα ζητήματα στο επίπεδο του ΠΟΕ. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα θα ήθελα να θέσω Ε, ισχύει το ότι έχετε ήδη μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κίνα. Έχετε πολύ στενές σχέσεις με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Από την εμπειρία σας στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα, θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα. Γιατί γεωγραφικά εσείς είσαστε τόσο πιο κοντά στην Κίνα που θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τις απόψεις γιατί από εντελώς διαφορετική γεωπολιτική πλευρά ε, μπορούμε να ακούσουμε τις εμπειρίες ενός ε, κράτους που έχει πολύ παρόμοιες αξίες με τις δικές μας. Και ε, ε, χαίρομαι που μιλήσατε κύριε Γκόφ για την ε, επέτειο της εκεχηρίας αυτή την εποχή τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ε, είναι θετικό το ότι ακούσαμε δύο λόγια και για τη διαδικασία της ειρήνης. Ευχαριστώ πολύ. Bern. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπέρναντ Λάγκε. Ακούσαμε ε, τα κοινά στοιχεία μεταξύ των λαών μας ε, ε, και είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι δεν έχουμε στοιχεία διαμάχης. Βλέπουμε στην άλλη άκρη του κόσμου μια χώρα που έχει ίδιες αξίες με τις δικές μας και με την οποία μπορούμε να έχουμε θετικές εμπορικές σχέσεις και χαίρομαι που ακούσα και εσά να αναφέρετε τις θετικέ σα εμπειρίες και να τονίζετε τα θετικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μιλήσαμε για τις διμερείς συμφωνίες που έχετε συνάψει. Το επενδυτικό κομμάτι αυτών των συμφωνιών ε, είναι ενδιαφέρον. Γνωρίζω ότι η Αυστραλία έχει δυσκολίες να συνάψει εμπορικές συμφωνίες και υπάρχουν ε, προβλήματα εθνικής κυριαρχίας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν και για τη Νέα Ζηλανδία προβλήματα σε τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες. Και όσον αφορά την επίλυση των διαφορών, έχετε να σχολιάσετε κάτι για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ, Μπέρντ, η κυρία Ντεσάνης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ακούμε. Έχουμε κοινέ αξίες και εξάγεται πολύ και σε εμά ε, γεωργικά προϊόντα πάνω απ' όλα. Χαμογελώντας το λέω ότι είναι πολύ καλό το κρέας που εξάγεται, αλλά και το δικό μας το γαλλικό είναι πολύ καλό επίσης. Ε, και δεν είναι, δεν είναι δεν είναι αστιάκι αυτό. Δύο σημεία να εξετάσουμε μαζί Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Κίνα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα υποτίμηση του κινέζικου νομίσματος και τις εξαγωγές σας που αυξάνονται με την Κίνα, οι εισαγωγές σας και Κίνες αυξάνονται. Μήπως κάτι μπορείτε να προσθέσετε για τις σχέσεις σας με την Κίνα, με ενδιαφέρει. Ευρύτερο το επόμενο ερώτημα. Είσαστε σε γεωγραφική περιοχή του κόσμου που περισσότερη επαφή έχετε με δημιουργία πλούτου, ανάπτυξη περισσότερο από ό,τι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προοπτικές σας οικονομικές της ανάπτυξης ποιες ήταν και πώς βλέπετε, πώς ατενίζετε την Ευρώπη, προς την Ευρώπη από εκεί που βρίσκεστε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τρεις ακόμη ομιλητές έχουμε. Πολ Μέρφι, Ντεμέντες και David Μάρτιν. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών γιατί θέλω να δώσω και στους προσκεκλημένους μας τη δυνατότητα να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Πολ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Ε, μπορεί να γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από, μερικές, ε, από μερικούς ε, μήνες καταψήφισε την άκτα μετά από διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπεγράφησαν πολλές αναφορές λόγω της καταπάτησης ελευθερίας του ίντερνετ και του λόγου. Η Νέα Ζηλανδία έχει, την, έχει, την έχει υπογράψει ε, την ε, συμφωνία αυτή. Χρειάζεται έξι ε, υπογραφές. Δεν την έχει βέβαια επικυρώσει ακόμα. Πρέπει να περάσει και από την ολόκληρη διαδικασία διαβούλευσης πριν επικυρωθεί. Αλλά το ερώτημά μου είναι πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη συμφωνία αυτή. το Μόσπονδο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας ε, πρότεινε να μην ε, επικυρωθεί γιατί μπορεί να υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα και μεγάλο κόστος από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ποια είναι η δική σας άποψη ε, και θα ήθελα να, να τοποθετηθείτε πριν ψηφίσετε, υπερψηφίσετε ή καταψηφίσετε. Όσον αφορά τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων που θα γίνει στο Όκλαντ συγκεκριμένα, θα ήθελα δύο πράγματα να ρωτήσω. Πρώτον, καταρχά, σε σχέση με τη διαδικασία, υπάρχουν πολλέ επικρίσει όσον αφορά τι διαπραγματεύσει του TPPA, όπω έγιναν και ε, με την άκτα, ότι είναι μυστικέ, ότι δεν υπάρχει δημόσια διαβούλευση, ότι δεν υπάρχει δημοσίευση των εγγράφων και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια πραγματική δημοκρατική συζήτηση όταν δεν συμμετέχει ο κόσμο, ότι πρέπει τέλο πάντων απλώ να βασιζόμαστε σε έγγραφα ποια είναι η άποψή σας για τη διαδικασία αυτή και ως προς το περιεχόμενο υπήρξαν ανησυχήσεις ε, από συνδικάτα και την κοινωνία των πολιτών για κάποια ζητήματα τα οποία γνωρίζουμε και εμείς εδώ ε, οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών ε, των επενδυτών που μπορεί να ευνοούν τα δικαιώματα των επενδυτών σε σχέση με τα δικαιώματα των συνδικάτων για των καταναλωτών ή ε, ας πούμε υπόθαλψη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κάτι ακόμη η απειλή για τις υπηρεσίες διαχείρισης των φαρμακευτικών, ε, για την ύπαρξη χαμηλών ε, τιμών φαρμάκων στη Νέα Ζηλανδία και ότι υπάρχει ανησυχία ότι η TPPA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδυναμώσει την ε, άποψη κατά των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Δεμέντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω σύντομα στους συναδέλφους μας βουλευτές. Είμαι μέλος της Επιτροπής της Αντιπροσωπείας για την Κίνα και για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Και πριν από δύο μέρες επέστρεψα από το Πεκίνο και Κατά την άποψή σα, μπορεί να υπάρξει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στι θέσει τη Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για το άνοιγμα προ την Ασία. Η Αυστραλίνη κυβέρνηση μόλις δημοσίευσε ένα πολύ σημαντικό ενδεικτικό έγγραφο. Η Αυστραλία ακριβώ σε αυτόν τον αιώνα και μέσω δηλώσεων ε, του κόμματος και του κράτους στον επίσημο τύπο στην Κίνα λένε ότι υπάρχει ένα πλήρες άνοιγμα της Αυστραλίας προς την Κίνα, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και οικονομικό, δημοσιονομικό και πολιτιστικό και πολιτικό. Δηλαδή έτσι το ερμηνεύουν στην Κίνα, ότι η Αυστραλία ανοίγεται πλήρως προς την Κίνα και αντί για την ε, γυραιά Ευρώπη. Και να το πούμε, αυτή τη στιγμή η κατάστασή μας δεν είναι και τόσο καλή. Τι έγινε, υπάρχει, συντάχθηκε ένα παρόμοιο κείμενο και πώς το βλέπετε το πράγμα έτσι, αυτό έτσι, έχει κατάσταση πλήρες άνοιγμα προς την Κίνα. Ευχαριστώ τελευταίο ομιλητή David Martin. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε χρόνο. Θα είμαι σύντομο. Καταρχά, ότι είναι φόρος τιμής ε, στην ικανότητα της ε, Νέας Ζηλανδίας ε, να πλασάρει τον εαυτό της ως χώρα τη ΑΣΕΑΝ όταν λέει ότι το Όκλαντ που είναι τόσο μακριά από την Ευρώπη είναι πολύ κοντά παρόλα αυτά στην Ευρώπη ενώ είναι πολύ πιο κοντά στο Πεκίνο. Τέλο πάντων πολύ καλό το marketing σα πρέπει να σα συγχαρώ. Δεύτερον, εγώ συμφωνώ με την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε πάρα πολύ ανοιχτή αγορά, τα επιθετικά σας συμφέροντα είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα είναι πολύ πιο ανοιχτή η αγορά σας για τα γεωργικά προϊόντα, η αγορά που θα έχετε για τα γεωργικά προϊόντα, αλλά τι μπορείτε εσείς αντάλλαγμα να δώσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μας προσελκύσετε σε διαπραγματεύσεις, γιατί να είμαστε και ειλικρινεί σε έναν εμπορικό κόσμο, πρέπει να έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν μπει σε διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία να έχει και κάποιο ε, Κάτι ακόμη θα ήθελα να ακούσω ε, από σας ε, Κάποιοι ήταν μέσα στη Γενέβη πριν από τέσσερα χρόνια, όπως εσύ. Εγώ μου ήμουν, εμείς, εγώ ήμουν έξω και θα ήθελα να μας πεις ε, μια ικανοποιητική εξήγηση για το τι δεν πήγε καλά, γιατί δεν πολύ καταλάβαμε και ποτέ. Νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη ερώτηση. Τελευταία και εγώ θα την έθετα, αλλά με πρόλαβες. Νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε σε 10 λεπτά να ακούσουμε και τι απαντήσει, ε, Ο Τζον Χέις. Ναι, βεβαίω, θα τα πω έτσι λίγο γρήγορα. Και μετά θα δώσω το στο συνάδελφο Γκόφ. Συγγνώμη, δεν γνωρίζω τα ονόματά σας ε, για την κυρία που ρώτησε για την Κίνα. 12 ώρες κάνουμε να πάμε στην Κίνα και 24 ώρες να πάμε στο Λονδίνο. Τόσο κοντά στην Κίνα δεν είμαστε, αυτό θέλω να πω. Το δικό μας ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι, είμαστε 4 εκατομμύρια άτομα. Η οικονομία δεν είναι απειλή για κανέναν. Ε, η αξία για τους Κινέζους είναι ότι υπήρξε ε, η πρακτική μιας πραγματικής ε, οικονομικής και εμπορικής σχέσης με έναν εταίρο που θα ήταν σοβαρός. Το πραγματικό όφελος για μας κατά τα τελευταία τρία χρόνια είναι οι εξαγωγές στην Κίνα. 3-4 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η αύξηση ετήσια του εμπορίου μας με την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε πολιτικός θέλει να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Το ερώτημα τώρα για τις εμπορικές μας σχέσεις. Έχουμε τελείω ανοιχτή επενδυτική πολιτική. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να επενδύσει στη Νέα Ζηλανδία, γιατί δεν έχουμε κεφάλαιο. Έχουμε μια οικονομία που είναι πέρα από την εμβέλεια της πολιτικής ε, και έχουμε και το θέμα της συναλλαγματικής ισοτιμίας που γίνεται σε επίπεδο κεντρικής τράπεζας ε, με κάποιο έλεγχο του πληθωρισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλει κανείς να αγοράσει γη στη Νέα Ζηλανδία ή αν θέλει να πάρει πάνω από 25% μετοχές σε μια εταιρεία πρέπει να περάσει από μια διαδικασία που λέγεται, από ένα τέλο πάντων γραφείο που λέγεται Γραφείο Εξωτερικών Επενδύσεων Overseas Investment Office και βλέπουν κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα. Να σας μιλώντας τώρα ως πολιτικός, αυτό, είναι, αυτό σημαίνει το εξής, ότι έρχονται οι Κινέζοι να αγοράσουν ε, εκτάσεις ε, ε, παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν μπορούσα εγώ τον James Cameron ή έναν Καναδό να τον εμποδίσω, ούτε κάποιον Ελβετό, κάποιον Αμερικάνο που έχει τη βάση του στην Ελβετία να έρθει να αγοράσει οτιδήποτε. Εννο, εννοώ ότι υπάρχει μια κάπως εσωτερική ξενοφοβία για να το πω έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι ισχύει η νομοθεσία που έχουμε ε, ε, στη χώρα μας ε, και από εκεί και πέρα τις 16 προτάσεις που μπορεί να είχαμε για αγορές τις εξετάζαμε κατά περίπτωση ανάλογα με το, κατα... με το πόσο μεγάλη αξία είχαν. τώρα το θέμα των εμπορικών σχέσεών μας με την Κίνα που προέκυψε πολλές φορές. Αν κάποιον τον κλέψει ένας Κινέζος δεν υπήρχε βάση ε, συναλλαγής μαζί του. Κάθε χρόνο τώρα μπορούμε να έχουμε τη βάση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου και νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική εμπορική εξέλιξη. Επίσης, και το λέω και εγώ εκπροσωπώντας τους δικούς μου ε, ψηφοφόρους, ότι η συμφωνία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να έχουν συναλλαγές με Κινέζους επιχειρηματίες, έχουν ε, τετραπλασιάσει και πενταπλασιάσει τις συναλλαγές τους, ε, συνεργάζονται καλά με τους Κινέζους και αυτές είναι βέβαια διαδικασίες ε, βοηθούν τις επιχειρήσεις με τέτοιο τρόπο που όταν εμείς συνήψαμε τη συμφωνία δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε καν. Το ερώτημα Ε, για την εξωτερική βοήθεια δεν το θυμάμαι, δεν το κατάλαβα πολύ καλά, οπότε θα το προσπεράσω. Για την άκτα και το TPP. Αυτές οι συμφωνίες από διαδικαστικής απόψεως στη Νέα Ζηλανδία θα τύχουν διαπραγμάτευσης από τους εμπορικούς διαπραγματευτές ε, υπό την ηγεσία των Υπουργών της κυβέρνησης και από καιρού εις καιρών και η δική μας Επιτροπή ενημερώνεται για το τι γίνεται. Υπάρχει τέλος πάντων κάποιο είδους παρακολούθηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει διαπραγμάτευση μιας εμπορικής συμφωνίας ε, από μια Επιτροπή σαν τη δική μας. Και εμείς επικρίνουμε τον τρόπο, ε, επικρίνουμε όπως επικρίνετε κι εσείς. Νομίζω όμως ότι η διαδικασία είναι ακέραιη, Παρακολουθείτε, ελέγχετε από την Επιτροπή μας, την Επιτροπή μου. Και τι διαφορά μπορεί να κάνει. Για παράδειγμα, είχαμε με τη Μαλαισία πρόσφατα μία συμφωνία που την υπογράψαμε. Όταν εμείς μπορούμε, μπορούμε να, μπορεί να γίνει αγορά στη Νέα Ζηλανδία 100% μιας εταιρεία από τη Μαλαισία, αλλά εμείς μπορούμε να αγοράσουμε μόνο 70% στην Μαλαισία. Αυτό δεν σημαίνει αμοιβαιότητα. Επίσης, μας ρωτήσατε για το Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Έχουμε ξεπεράσει τους Αυστραλούς σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους Κινέζους παρά το γεγονός ότι είμαστε τόσο μακριά, είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον. Αν εμείς σταματήσουμε να αγοράζουμε από την Κίνα και μετά η Κίνα σταματήσει να αγοράζει από την Αυστραλία άνθρακα και άλλα προϊόντα, τότε οι Αυστραλοί θα σταματήσουν να αγοράζουν προϊόντα από εμά. Και εμεί είμαστε, η μεγαλ... για μας είναι αυτή η μεγαλύτερη αγορά. Δηλαδή, ο ένα τερνίζεται και ο άλλο έχει πρόβλημα. Καταλαβαίνετε πόσο, δεμέν, πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε. και κάνατε και μία ερώτηση για το σε τι είναι επικερδές αυτό για την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να εκφοβίζουμε τον κόσμο με την ακαιρεότητα. Αν μπορούμε να έχουμε μια, ελεύθερη, μια, μια, μια συμφωνία ελεύθερη, δεδομένων των αξιών ε, που έχουμε, εσείς συναλλάσσεστε μαζί, μαζί μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία του Κοινοβουλίου ε, σε μια ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ Νέας Ζηλανδία και Ευρωπαϊκής Ένωση. Γι' αυτό είμαστε εδώ και όχι κάπου αλλού και θα, το, θα ξανάρθουμε και πολλές φορές να το πούμε αυτό. Θα μας ξαναδείτε. Και ελπίζουμε σύντομα σύντομα σε ευρωπαϊκό χρόνο λέω, να τα καταφέρουμε. Γιατί είμαστε μία από τις εννέα μόνο χώρες που σε μη προτιμησιακές τιμές πουλάει σε αυτή την αγορά. Μπορείτε να μας, ε, να μας ζητήσετε ε, δασμούς, αλλά πρέπει να αναρωτηθείτε για ποιο, σε τι θα χρησιμεύσουν. Με ρωτήσατε γιατί το πράσινο δωμάτιο απέτυχε στη Γενέβη. Ξέρετε ότι η πολιτική βασίζεται στο συμβιβασμό και η θέληση συμβιβασμού για ένα συλλογικό το πρόβλημα με το να γίνει μία αλλαγή είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν συμφέρον ε, ε, να, να, ισχύσει η παλαιά πολιτική θα αγωνιστούν με νύχια και με δόντια να την κρατήσουν και όσοι είναι υπέρμαχοι της ε, ε επόμενης της, της αλλαγής πάλι θα αγωνιστούν και δεν υπάρχει συμβασμός γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν συμφέροντα για συγκεκριμένους τομείς, ε, ακόμη και αν είναι ένας αυτός ο τομέας και ακόμη και κάποιος να αντιστέκεται, δεν προχωράει η συμφωνία. διότι το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τις ασιατικές χώρες δεν σημαίνει για παράδειγμα ότι απομακρυνόμαστε από τους παραδοσιακούς μας φίλους και συμμάχους. Και το λέω αυτό λόγω του διπολικού κόσμου, οι Ηνωμένε Πολιτείε Κίνα. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εκεί, να ασκεί την επιρροή της ε, ευρύτερα για να μπορέσει να εξισορροπεί τα συμφέροντα αυτών των δύο μεγάλων ε, ε, υπερδυνάμεων. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση και επειδή ο Πολ έθεσε αυτή την ερώτηση την τελευταία, ναι, είναι σημαντικό να έχει κανείς ένα, ένα, ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτών, ε, γιατί εσύ μπορεί να έχεις αυτόν τον κανόνα και να έχεις και κράτος δικαίου, αλλά η άλλη χώρα μπορεί να μην έχει το κράτος δικαίου κατά την ίδια έννοια και πρέπει να δει κανείς με ποιους ε, συναλλάσσεται. Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση για το TPPA, για παράδειγμα, πρέπει να ληφθεί υπόψη το κυρίαρχο δικαίωμα της κάθε, της κάθε να νομοθετεί, να ρυθμίζει για το κοινό καλό, για την υγεία και το περιβάλλον και εμείς δεν πρόκειται να αποποιηθούμε αυτού του δικαιώματος. Συγγνώμη για τις ερωτήσεις που δεν απαντήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Right. <clears throat> Well, on behalf of you all, I'd like to... Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων τους προσκεκλημένους μας από τη Νέα Ζηλανδία και τους προσκεκλημένους και τον πρέσβη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση όπως μας αρέσει να έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας. Uh, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, έχετε έτοιμες τις κάρτε σας για την ψηφοφορία. Αν δεν έχετε την κάρτα σας, παρακαλώ να μας το πείτε, να μας πείτε τι ψηφίζετε κάθε φορά. Ζητώ συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Τώρα θα ξεκινήσουμε όμως την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σημείο 14 εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής. Όπως θα θυμάστε, στις 11 Οκτωβρίου κάναμε μια ενδεικτική ψηφοφορία ε, για τις ε, δύο διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου σχετικά με τις συμφωνίες ε, Κεντρική Αμερική, Κολομβία και Περού. Και τώρα φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία για την συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την εφαρμογή των διμερών ρητρών διασφάλισης και το μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες. Μετά από δύο άτυπες διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου με την Κορεπέρ εγκρίθηκε η συμφωνία. Η Κορεπέρ στις 31 Οκτωβρίου ενέκρινε το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχουν τρεις επιφυλάξεις στο Συμβούλιο, αλλά αναμένεται ότι θα αρθούν οι επιφυλάξεις σύντομα πριν από την ψήφο στην Ολομέλεια, το κείμενο, ε, ελπίζουμε, ε, ε, πριν από την συζήτηση στην Ολομέλεια, ελπίζουμε ότι θα έχουν αρθεί οι επιφυλάξει. Σα έχει μοιραστεί το κείμενο και θα ήθελα να υποφεληθώ τη ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον εισηγητή που δεν είναι παρόν, τον Γιώργο Λάικφριντ και τον κύριο Μπέντ Λάγκε. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. There is only one vote. It will θα γίνει μόνο μία ψηφοφορία, η τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. No... Εψήφισαν όλοι. Εσείς δεν έχετε κάρτα. Το σημειώνουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 in favor, uh, two against and three abstentions. Plus one. Oh, plus one. So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 19 ψήφοι, 20, 20 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 3 αποχές. Για το σημείο 15. Σημείο 16. χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις ως υποστήριξη έναντι της παγκοσμιοποίησης. Γιάν Ζαραντήλ. Είστε έτοιμοι. Συμβαστική τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Περνάμε στην 24 του Πολ Μέρφυ υπέρ. Μάλλον θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία γι' αυτό. Θα το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 44 και 25 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Συμφωνείτε ή όχι. Α, δεν ξέρετε. Απέχετε. Απερίφθη. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεδραστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 33 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Καταπίπτει. Άρα περνάμε στην τροπολογία 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, καταπίπτει. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, απο... Α, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Και εδώ πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 καταπίπτει 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ. Είναι σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές. Πάλι θα πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν μπορούσα να το κρίνω. Δεν βλέπω ότι ψηφίζει το ΕΛΚ. Για τη 19 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Με ναι, ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε μετά τις τροποποιήσεις. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. 17. Yeah. Just one vote, isn't it? Oh, do I? now come to a vote on the draft recommendation. Σχέδιο σύσταση δεύτερη ανάγνωση για την περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδότηση στη Γεωργία. Επανεπισημαίνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, δεν υπήρξαν άλλες τροπολογίες, ε, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικός, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, το κείμενο στο σύνολό του, το κείμενο στο σύνολό του, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται ψηφοφορία, πέρας. 23 υπέρ, 1 ε, κατά και 2 αποχές. Περνάμε τώρα στο σημείο 18. Ψηφοφορία για την ε, για την έκθεση Σούστα. Έχουν συμπεριληφθεί κάποιες ψηφοφορίες. Πρώτη ψηφοφορία, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Υπέρ και πάλι σηκώστε καλά τα χέρια. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. 15 υπέρ 11 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλό θα ήταν να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν καταλαβαίνω πώς ψηφίζει το ΕΛΚ. Υπέρ. Παρακαλώ σηκώντε καλά τα χεράκια. Υπέρ. Κατά. Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Έναρξη επιφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ 11 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Και οι 5 μαζί τις ψηφίζουμε. 5 και 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 19, 19. 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 20 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Κατά τμήματα ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. κατά πίπτη. Τροπολογία 1. Και 7 μαζί. Υπέρ. καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο τμήμα. 23 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 και 7 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομοφόνο συγχαρητήρια κύριε Σιγητά 19, 19. Uh, συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Ιράκ. Γνωμοδότηση σε σχέση με τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ. Κρίμα που είναι μόνο γνωμοδότηση η έκθεσή μα, διότι πρόκειται για μια πλήρη εμπορική συμφωνία με συμβατότητα ΠΟΕ και μάλιστα με συμβατότητα με το μηχανισμό επίλυσης του ΠΟΕ. Ο κύριος Μέντες ήταν ο αρχικός εισηγητής. Ήταν στην Επιτροπή, αλλά δεν είναι πια μέλος της Επιτροπής μας. Μαρία Μπαντία είναι τώρα η συγγήτρια που αποφάσισε να διατηρήσει την αρχική θέση του εισηγητή και επομένως να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. The is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 21, ψηφί 21 ψήφοι υπέρ, 3 ε, ψήφοι κατά και δύο αποχές. Yeah. Uh, yeah. Thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην ακρόαση. Okay. Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, η δημόσια ακρόασή μας αφορά την επενδυτική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωσης Κίνα. Ακούσαμε λίγο από τη Νέα Ζηλανδία και την αντιπροσωπεία της πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Επειδή υπάρχουν διμερείς σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνας πριν από 37, εδώ και 37 χρόνια έχουν ε, επεκταθεί από 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε το 78 σε 448 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011. Είναι καταπληκτική η αύξηση. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν φεύγετε, να φεύγετε ήσυχα. Καταλαβαίνω ότι μετά την ψηφοφορία θέλετε να φύγετε, αλλά παρακαλώ λίγη ησυχία. Λοιπόν, από 4 δισεκατομμύρια του 78 φτάσαμε σε 488 το 2011 είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγαλύτερος αποδέκτης εξαγωγών ε, και ε, δεύτερος εταίρος μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, ε, το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 292 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε αγαθά, 17% από την Κίνα των εισαγωγών και οι εξαγωγές ε, είναι όγκου 123 δις ευρώ στην Κίνα το 2011. Είναι μία από τις ε, πρώτες πέντε πηγές άμεσων ξένων επενδύσεων, 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 στην Κίνα. Αυξάνονται ραγδαία οι επενδύσεις από το 2009 και την κρίση, αλλά παραμένουν ε, σε μέτριο επίπεδο. 3,9 δις ε, ευρώ. Θα γνωρίζετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, θεωρεί ότι οι ξένες επενδύσεις είναι τμήμα των ε, ενωσιακών αρμοδιοτήτων δεδομένου, δεδομένης της διμερούς συμφωνίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα πολύ από τις, πολλές από τις νέες ελεύθερες συμφωνίες εμπορίου καλύπτουν όλο και περισσότερα ζητήματα ε, και επενδυτικά θέματα. Η Σύνοδος της Βρυξέλλες της 21 Νοεμβρίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας πρότεινε έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία επενδυτική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας ως συντομότερο δυνατόν με στόχο την προώθηση και διευκόλυνση ε, των επενδύσεων ε, και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ε. Θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές όλους τους τομείς ε, ενδιαφέροντος και για τις δύο τιμές, με την επιφύλαξη βέβαια του τελικού αποτελέσματος. Επίσης αποφάσισαν ενίσχυση τεχνικών συζητήσεων προπαρασκευαστικών για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή μας θέλει να συμβάλλει οργανώνοντας αυτήν την επίκαιρη ακρόαση. Σήμερα ε, τα μέλη του πάνελ μας θα συζητήσουν για τα ενδεχόμενα εμπόδια αλλά και τα ωφέλη μιας τέτοιας ε, συμφωνίας. Ε, να δούμε ποια είναι η κατάσταση μεταξύ των... η κατάσταση σαν ξένες επενδύσεις Δύο πάνελ θα έχουμε στην ακρόασή μας. Μετά από την παρουσίαση των μελών του πάνελ, καλό είναι να υπάρξουν δύο γύροι ερωτήσεων και μετά απαντήσεις και σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, η εμπορική αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχει επίσης προσκληθεί να σχολιάσει. Λοιπόν, να δώσω το λόγο τρεις, για τρία λεπτά στον κύριο Ραβελίνο πρόεδρο της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Κύριε Ραβελίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου προσφέρετε τη δυνατότητα να κάνω μια εισήγηση για την αποστολή μας η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο μας πέρασε πριν από δύο μέρες, ε, τρεις ε, η αντιπροσωπεία μας με την Κίνα για 34η συνάντηση Ευρώπης-Κίνας πήγαμε στην Κίνα ακριβώς και είμαστε η τελευταία επίσημη αντιπροσωπεία η οποία μετέβη στο Πεκίνο πριν από το συνέδριο του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Πέρα από μια τεχνική εισήγηση θα πρέπει να είναι και πολιτική εισήγηση για το τι αποκομίσαμε σαν εντυπώσεις, τι βρήκαμε, τι συναντήσαμε, ποιες προοπτικές υπάρχουν στην Κίνα. Τα στοιχεία σχέσεως μεταξύ των δύο το 2011 430 δισεκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια παραπάνω από ότι το 2010. Οι άμεσε επενδύσει στην Κίνα το 2010 ήταν 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία. Νομίζω ότι καθηγητές πανεπιστημιακοί που θα λάβουν το λόγο μετά από μένα θα μπορούν αυτά να σας τα εξηγήσουν τα τεχνικά στοιχεία καλύτερα σαν πρόεδρος της πολιτικής αντιπροσωπείας η οποία επισκέφτηκε την Κίνα θα ήθελα να σας ε, μεταβιβάσω τις εντυπώσεις μου. Πρώτα απ' όλα, πρώτη εντύπωση, απεσιοδοξία στις επίσημες συναντήσεις που είχαμε με το Γενικό Διευθυντή Διοικητή της ε, Bank of China που μας υποδέχτηκε και ακούσαμε για το πώς έχουν οι επενδύσεις της Κίνας στην Ευρώπη. Μια κάποια απεσιοδοξία όσον αφορά την υγεία του ευρώ. Αυτή εμφανίστηκε καθαρά, εκφράστηκε καθαρά με διστάζουν ε, απόλυτα και πιστεύουν ότι θα πρέπει να περιμένουν να περιμένουν μέχρι να έρθει η στιγμή να συνεχίσουν να επενδύουν στην Ήπειρό μας. Δισταγμός λοιπόν. Δεύτερο, η Κίνα ακόμα σήμερα αποτελεί πάντως μια τεράστια δυνατότητα γιατί Πεκίνο, Σανγκάι, στις κύριες μεγαλύτερες πόλεις υπάρχει μια διάθεση για επένδυση για αγορές προϊόντων της Ευρώπης. Ο ιός της κατανάλωσης έφτασε και στην Κίνα και έφτασε από την Ευρώπη. Η πρώτη μας εκτίμηση από τη στιγμή που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο είναι ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα στο Πεκίνο ήταν αυτοκίνητα πολυτελή ευρωπαϊκά, Φεράρι και Mercedes, πολλές στο Πεκίνο. Και αυτή είναι μια εκτίμηση που μας κάνει να θεωρούμε ότι το μέσο επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς ε, του Κινέζου πολίτη και υπάρχει η διάθεση από πλευράς του να αγοράσει αγαθά κινέζικα. Ε, στο Λουί Βουητών ε, επισκεφθήκαμε καταστήματα με τρομερό κύκλο εργασιών όπως και οι γερμανικές τεχνολογικές εταιρείες η Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία σε αυτήν την Κίνα, την αστική της, του Πεκίνου και της Σανγκάης. Εκεί εμφανίζεται η ευμάρια και η ευμάρια εκφράζεται με δυτικό τρόπο αγορών και στις επαρχίες. Πήγαμε και στην πόλη Τσόντσινγκ στο Λουμπέι στην επαρχία και είδαμε την Ήπεθρο. Τι διαπιστώσαμε. Όλο και περισσότερες οικοδομές, κτίρια, πολύ σημαντικές επενδύσεις στη Σοντσίνγκ που από το 1996 και μετά προσέχτηκε ιδιαίτερα από την κινέζικη κυβέρνηση για μια δημογραφική τρομερή ανάπτυξη το σύνολο το γεωγραφικό της περιοχής εκεί στο Σοντζίνγκ είναι περίπου 40 εκατομμύρια κάτοικοι ενώ ο κεντρικός πυρήνας της πόλης ε, είναι το κέντρο της πόλης έχει περίπου 13 εκατομμύρια κατοίκους. Σονζίνγκ εκεί γίνονται τρομερές επενδύσεις ε, κατασκευάζουν παντού και στο κέντρο και θα έχουν και ένα αεροδρόμιο του χρόνου με τέσσερις διαδρόμους προσγείωσης με 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες το χρόνο και έχουν προγραμματίσει την πόλη με κατοικίες ε, τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα, τι θα γίνει με την υψηλή τεχνολογία. Να μία πόλη ακόμα που μέσα σε πέντε χρόνια το κέντρο, μάλλον ε, η περιοχή αυτή παραγωγής θα έχει 2,5 εκατομμύρια κατοίκους. Απαιτούνται επενδύσεις στην Κίνα και στις επαρχίες υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Αυτός ο πολυάριθμος λαός, πολυπληθής λαός θα μπορούσε να προσφέρει μία ελπίδα στην Ευρώπη που ταλανίζεται από την κρίση. Αλλά τι μας είπαν οι Κινέζοι συνάδελφοι, οι βουλευτές οι Κινέζοι από την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις προοπτικές του του συνεδρίου του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος μας έκανε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε και άλλους τομείς. Τις 8 Νοεμβρίου που θα ξεκινήσει αυτό το συνέδριο θα δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι Κινέζοι μια διαφορετική ποιότητα ζωής δηλαδή με επενδύσει στον τομέα της υγείας και οι δημόσιοι υπάλληλοι των μεγάλων πόλεων σε πέντε χρόνια θα πρέπει πρέπει να έχουν ε, υγειονομική ασφάλιση δωρεάν και από κοινωνικής πλευράς θα υπάρξει φροντίδα ε, για τους συλλοκιωμένους και για τους ανίκανους προς εργασία και μια δημιουργική ανάπτυξη στον κοινωνικό τομέα. Στη συνάντηση αυτή θα μπορούσαμε να δούμε και άλλες δυνατότητες επένδυσης πέρα από τα αιτήματα των Κινέζων φίλων μας οικονομία αγοράς, οι δυνατότητες να απαλληφθούν οι δασμοί, το εμπάργκο το στρατιωτικό και τα συνηθισμένα που γνωρίζετε όλοι σας καλύτερα από μένα και πώς θα δούμε ένα σύνορο με μια ισορροπημένη βοήθεια. Σας παρακαλώ μήπως θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε γιατί ότι δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, εντάξει, θα ολοκληρώσω αμέσως. Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω σε λεπτομέρειες αυτό τον καινοτόμο τομέα της υγείας που ανοίγει αγορές στην Κίνα που έχουμε εμεί το know-how στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να επενδύσουμε και στον τομέα αυτό στην Κίνα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε ότι θα σας παρουσιάσω τους ε, συμμετέχοντες. Ο καθηγητής Ντάνιελ Βαντεμπούκα από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας ήταν διευθυντής μέχρι το 1996 και πρόεδρος του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Πολιτικής και Διοίκησης από το 1996 μέχρι το 2000. Ήταν ακαδημαϊκός ε, διευθυντής του Κέντρου Ευρώπης-Κίνας στη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας μέχρι το 2002 και τώρα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει γράψει πολλά βιβλία για θέματα ξένων επενδύσεων και ξένων άμεσων επενδύσεων και είναι εμπειρογνώμων σε πολλά θέματα επενδύσεων στην Κίνα. Ασχολήθηκε με προγράμματα έρευνας για το Βελγικό κράτος, για το Βελγικό Υπουργείο Οικονομικών και για τα Ηνωμένα Έθνη. Για τον ΟΣΑ, το, Ευρωπαϊκό, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς. Ο δεύτερος προσκεκλημένος μας είναι ο καθηγητής κύριος Χάι Γιάν Τζάνγκ, πάλι από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, από το, τη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας. Έχει διδακτορικό σε θέματα δημόσιας διοίκησης από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Επίσης είναι επισκέπτης καθηγητής σε πολλά κινέζικα πανεπιστήμια και διδάσκει σε διεθνή προγράμματα MBA για τις ασιατικές επιχειρήσεις, για το περιβάλλον και για τη στρατηγική διαχείριση. Ενδιαφέρεται για θέματα όπως οι διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες για τις επενδύσεις και για τις επιχειρήσεις στην Κίνα και στο εξωτερικό, άμεσες ξένες επενδύσεις και κοινοπραξίες και επενδύσεις σε μεταβατικές οικονομίες. Ο τρίτος προσκεκλημένος είναι ο κύριος Dirk Mons από το Εμπορικό Επιμελητήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, είναι ο Γενικός Γραμματέας από την 1η Μαρτίου του 2009. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του επιμελητηρίου σε ολόκληρη την Κίνα. Πριν αναλάβει αυτή τη θέση στο Επιμελητήριο Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, είχε ε, πολλές ε, θέσεις στην επιτυχή του σταδιοδρομία σε μια μεγάλη εταιρεία ε, ποτών με αρμοδιότητες για την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού και έχει ζήσει με την οικογένειά του στην Αφρία, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Ντάνιελ Μπούλκε πρώτα. Still Yeah. Άναψε το μικροφωνό μου. Ωραία. Δεν ξέρω τι να πω. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Το θέμα το σημερινό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και προσπαθώ να καλύψω 70 διαφάνειες σε 10 λεπτά, άρα θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Μην ανησυχείτε όμως τα περισσότερα είναι κυρίως ε, ιστορικό και θα μπορέσετε να τις δείτε αργότερα με την ησυχία σας ε, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Σύντομα να σας πω καταρχάς ε, σε σχέση με το καθεστώς της πολιτικής και την εξωστρεφή άμεση επένδυση της Κίνας. Ε, ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε μία σύντομη σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι πιο ανεπτυγμένες χώρες όπου πολλές κινέζικες επενδύσεις ε, καταλήγουν σήμερα. Θα προσπαθήσω επίσης να παρουσιάσω μία πιο πλήρη εικόνα, γιατί οι συνάδελφοί μου και εγώ ε, όταν ε, εκπονήσαμε τη μελέτη έχουμε λίγο διαφορετική προοπτική σε σχέση με τις υπόλοιπες μελέτες. Χρησιμοποιήσαμε πολύ ευρύτερα δεδομένα πολύ περισσότερα δεδομένα. Ε, θα προσπαθήσω επίσης να αναφερθώ σε, κάποια, σε κάποιες ανησυχίες. Δέκα λεπτά έχω στη διάθεσή μου, το ξέρω, δεν καταφέρω να τα καλύψω όλα. Θα με διακόψει βεβαίως ο Πρόεδρος ε, και ενδεχομένως ε, να προκύψουν κάποια θέματα στη συζήτηση. Το θέμα της εσωστρεφούς και εξωστρεφούς ε, άμεσης ε, ξένης επένδυσης και των ροών της έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Η εξωστρεφής επένδυση προέκυψε πολύ αργότερα με, με μετά το μέσο της προηγούμενης ε, δεκαετίας και μου αρέσει πολύ αυτό που έγραψε το, Fortune, το περιοδικό Fortune το 2009 το 2009 εξακολουθεί όμως να ισχύει και μάλιστα όλο και περισσότερο για την κατάσταση στην ε, Ευρώπη και όχι μόνο στη ΣΥΠΑ. Εδώ έχουμε μια γραφική παράσταση που μας δείχνει από τη μία την ε, παγκόσμια εξωστρεφή επένδυση και από την άλλη την κινέζικη ε, στο εξωτερικό. Βλέπετε δηλαδή ότι είναι διαφορετικός ο όγκος αυτών των ροών, αλλά έχουμε αριστερά και δεξιά τα δύο, τις δύο παραστάσεις για να μπορείτε να, να τα συγκρίνεται και βλέπετε τα τελευταία δύο χρόνια, το, της κρίσης δηλαδή, ε, ότι υπήρξε μείωση ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά εξακολούθησε να αυξάνεται η οι κινέζικες επενδύσεις, σε κάτι το οποίο είναι ένα πολύ αξιέπαινο επίτευγμα. Εδώ βλέπετε τις έκροες, ε, οι επενδύσεις δηλαδή από την Κίνα στο εξωτερικό κατ' και είναι πραγματικά μια τεράστια αύξηση. Αν δει κανεί ε, τη σχέση μεταξύ 2006 και 2011, να μην σας πω 2012, έχει πενταπλασιαστεί τουλάχιστον, κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Ε, όσο, είναι, όσο μεγαλύτερες είναι οι ροές ετησίως, ε, βέβαια αυξάνονται και οι επιχειρήσεις, οι επενδύσεις που προσελκύεις. Το βλέπετε αυτό το 2011 έχει αυξηθεί σε 424 εκατομμύρια ε, δολάρια ε, Αμερικής. Να το δούμε αυτό σε σχέση με άλλους επενδυτές. Η Κίνα δεν είναι από τους μεγαλύτερους, όμως είναι ήδη πέμπτη στην ταξινόμηση του 2010. Και αν προσθέσει κανείς το Χονγκ Κόνγκ θα έφτανε στη δεύτερη θέση. Και βέβαια είναι αξιέπαινο ότι αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Ας δούμε και τους τομείς. Ε, συχνά ακούγεται ότι οι επενδύσεις αφορούν κυρίως ορυχεία, πετρέλαια, λιανικό εμπόριο. Βλέπετε όμως ότι και η μεταποίηση αυξάνεται όλο και περισσότερο. Το ποσοστό ανάπτυξης έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Γιατί, γιατί υπάρχει ένας ε, επαναπροσανατολισμός προς τις αναπτυσσόμενες χώρες της κινέσικης επενδύσης και εκεί γίνεται ιδιαίτερη μεταποίηση. Βλέπουμε τώρα μία προβολή του τι θα συμβεί στην κινέζικη επένδυση εάν συνεχίσει η παρούσα τάση. Το 2022 η Κίνα θα είναι η πιο, ο πιο σημαντικός εξωστρεφής επενδυτής παγκοσμίως, θα έχει ξεπεράσει και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Άλλες προβολές ε, αναφέρουν μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα ε, νούμερα και ότι μπορεί να συμβεί και νωρίτερα από το 2022. Μόνο 6% της συνολικής επένδυσης είναι η Ευρώπη ε, ως αποδέκτης των κινέζικων επενδύσεων ήταν ε, σε ίσο επίπεδο και χαμηλότερο από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αυξήσει το μερίδιό της. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τα κίνητρα των κινέζικων επενδύσεων σε γενικές γραμμές, όμως μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό είναι συγκρίσιμο με άλλους ξένους επενδυτές. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει όμως το εξής φαινόμενο. Οι επενδυτές ουσιαστικά αναζητούν ε, τεχνολογία στο εξωτερικό, ε, τεχνογνωσία, κάτι που τους, ε, που τους ενδιαφέρει, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στην ε, εσωτερική τους αγορά. Δεν θα μπω στις διάφορες, στα διάφορα είδη. Συμπερασματικά απλώ να πω ότι οι ακαδημαϊκοί, οι πανεπιστημιακοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα τη άμεση ξένη επένδυσης έχουν αποδεχθεί ότι κάπως πρέπει να προσαρμόσουμε τα πράγματα γιατί θεωρούσαμε ότι οι εταιρείε άμεσων ξένων επενδύσεων ε, ήταν εταιρείε που μπορούν να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα σε σχέση με τι τοπικέ εταιρείε που επενδύουν στο εξωτερικό. Εδώ έχουμε μια άλλη κατάσταση ε, χώρες που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες παρόλα αυτά πηγαίνουν στο εξωτερικό γιατί θέλουν ε, αυτές τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που ανέφερα. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ε, χαρακτηριστικό της Κίνας αυτή τη στιγμή. Για, πολιτική δεν θα μπω σε, για τις πολιτικές δεν θα μπω σε Από το 2000 όταν άρχισε αυτή η εξωστρεφής πολιτική έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επένδυση από την Κίνα και σύμφωνα με έρευνες από το CCPIT φαίνεται ότι οι εταιρείε επηρεάστηκαν από την κυβερνητική πολιτική να ε, δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Κάτι που επίσης θεωρώ ότι είναι δύσκολο και εξαιρετικό είναι ότι το 2006 η Κίνα ε, πολύ ανοιχτά ήθελε ξένες επενδύσεις. Δεν ξέρω πολλές χώρες όπου να έγιναν τέτοιες δηλώσεις, το διαβάζω πολύ γρήγορα. Θα υποστηρίξουμε ειδικευμένες επιχειρήσεις ε, που διαστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, θα, ε, ε, υπηρεσίες, δίκτυα υπηρεσιών, έρευνα και ανάπτυξη σε, άλλες χώρες. Και κατόπιν αυτού άρχισε μια τεράστια ανάπτυξη ε, των σχετικών πολιτικών και, των επενδύσεων εκτός Κίνας. Να σας πω για κάποιες εξαγορές που έγιναν. Έμαθα προσφάτως ότι 15 αμπελώνες ε, αγοράστηκαν από κινέζικες εταιρείες. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο αυτό. Volvo, Medion, ε, συνάδελφοι μπορεί να εμβαθύνουν σε αυτό. Πρόσφατα παραδείγματα, πολύ γρήγορα πάω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κάθε εβδομάδα αυξάνεται το κατάλογος γιατί όλο και περισσότερες κινέζικες εταιρείες ε, βάζουν πόδι στην Ευρώπη. Όπως βλέπετε από τη συγκεκριμένη γραφική, από τη συγκεκριμένη απεικόνηση, ε, η Ευρώπη έχει υποδεχθεί πάρα πολλές επενδύσεις από την Κίνα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, πολύ πιο ραγδαία από ό,τι άλλα μέρη του κόσμου. Δείτε και αυτή την πίτα. Ε, αυξάνεται πολύ γρήγορα ο ρυθμός, αλλά αν δει κανείς τα αποτελέσματα, το μερίδιο της, της Κίνας είναι 0,1-0,2% από τις συνολικές ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη. Και βεβαίως ε, αυτό επηρεάζεται από τις επενδύσεις ε, ε, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Κάποιοι θα, θα λέγανε, ας πούμε, ότι εφόσον αν, είναι, ανησυχείτε, αλλά ανησυχείτε για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό ακόμα. Ναι, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης ε, είναι πάρα πολύ ε, έντονος και συνεπώς πολύ ανησυχητικός. Δεν έχουμε χρόνο, προχωράω και πάλι πιο γρήγορα. Σας δίνω κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι Κινέζοι έχουν επενδύσει περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη από ότι στη Βόρεια Αμερική και στις Ηνωμένε Πολιτείες και πιστεύουμε ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις μπλόκαραν οι διαδικασίες ε, όχι από το CFIUS υποχρεωτικά, αλλά ε, και γιατί δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι είπαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Αυξάνεται λοιπόν το μερίδιο της Ευρώπης όπως είπα σε σχέση με τις εξαγορές. Δεν χρειάζεται να σας πείσω για όλα αυτά τα πράγματα οπότε τα προσπερνάω. Όλες αυτές οι μελέτες ε, εξετάζουν τους ισολογισμούς, τα σχετικά δεδομένα και τα ε, νούμερα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Όμως εμείς στη σχολή management στην Αμβέρσα είδαμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Ξεκινήσαμε από 18 εκατομμύρια περίπου εταιρείε ε, με έδρα την Ευρώπη, πρόκειται για τη βάση δεδομένων αμαντέους, 4.676 επιχειρήσει είναι κινέζικες, 28 ευρωπαϊκές χώρες και καταλήξαμε σε 4.525 κοινωνικές, ε, κινέζικες εταιρείες άμεσων ξένων επενδύσεων ή θηγατρικές τους. Οι επιχειρήσεις ήταν μικρές, οικογενειακού τύπου, επιχειρηματικού τύπου. Στις υπόλοιπε έρευνε αυτό δεν αναφέρεται καθόλου γιατί θεωρείται ένα διαφορετικό ξεχωριστό θέμα. 16% είναι, είναι ε, θηγατρικές μικρές ε, και χρησιμοποιώ τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και ε, εστιάζονται κυρίως και δεν, μην κοιτάτε αυτό το χάρτη γιατί αυτό είναι από μια ε, μελέτη προγενέστερη φαίνεται όμως ότι οι τρεις χώρες που προσελκύουν τις περισσότερες κινέζικες επενδύξεις είναι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο Εμεί όμω σας δείχνουμε αυτή τη χαρτογράφηση των κινέζικων επενδύσεων και βλέπετε ότι οι περισσότερες είναι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είναι όμως οι μικρέ, και επαναλαμβάνω, είναι μια διαφορετική οπτική γωνία αυτή. Οι βασικές, ε, η βασική εστίαση των κινέζικων επιχειρήσεων είναι Μόσχα, Βουδαπέστη, Βουκουρέστη, Αμβούργο, ε, Λονδίνο, Ντίσελντορφ, η Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, εκπροσωπείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, ε, λόγια ανησυχία τώρα. Αν είναι διαφορετική η εξωστρεφής ξένη επένδυση της Κίνας, από, της Κίνας από άλλες χώρες. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα στοιχείο σχεδιασμού. Μειώνεται, αλλά υπάρχει. Να σκεφτεί κανείς, ε, για παράδειγμα, την εστίαση σε διάφορους τομείς, ε, ο ρόλος των κρατικών επιχειρήσεων έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ είχε μειωθεί στο παρελθόν. Είναι πραγματικά μια μοναδική κατάσταση αυτή και υπάρχει και έντονη κυβερνητική υποστήριξη των εξωστρεφών επενδύσεων. Εγώ το, θεωρώ, το αναφέρω ως go αυτό, go out, βγείτε προς τα έξω δηλαδή. Και είναι αυτό που έκαναν άλλωστε οι κινέζικες εταιρείες για αύξηση του ενεργητικού του το κάνουν κυρίω. και υπάρχει μια έλλειψη ισορροπία μεταξύ τη προσέγγιση τη Κίνα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αμοιβαιότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πριν από μερικέ χώρε, μέρε, είδα ότι ο Καναδά προσπαθεί τουλάχιστον να συζητήσει αυτό το θέμα. Πρέπει να σταματήσω. Έχω κάποια επιχειρήματα, αλλά ενδεχομένω να προκύψουν στην ε, συζήτηση. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο γιατί πραγματικά αυτό που μας είπατε ήταν πολύ συναρπαστικό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα υπάρξουν ε, τεράστιες ευκαιρίες ε, για την Ευρώπη με τις κινέζικες επενδύσεις. Ε, επόμενος ομιλητής είναι... ο, κύριος, ο καθηγητής Χάιεν Ζάγκ Έχετε το λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω κάποιες πτυχές στα όσα παρουσίασε ο καθηγητής Ντάνιελ Βαντενμπούλκε από την Ευρωπαϊκή Προοπτική και από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην παρουσίασή μου υπάρχουν τέσσερα τμήματα τα βασικά γνωρίσματα των Κινέζων επενδυτών στην Ευρώπη. Θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένες περιπτώσεις για να δούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και τέλος ε, θα μιλήσω εν συντομία για την ε, πολιτική των κινέζικων επενδύσεων στην Ευρώπη. Ε, ας δούμε λοιπόν αν οι Κινέζοι επενδυτές είναι διαφορετικοί από τους προηγούμενους επενδυτές. Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι, γιατί δεν είναι καινούριο φαινόμενο αυτό. Ήδη τη δεκαετία του 60 υπήρχαν, υπήρχε η αμερικανική πρόκληση στην Ευρώπη και αργότερα είχαμε μια ιαπωνική επιχειρηματική επιδρομή στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτή τη φορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση γιατί οι επενδυτές προέρχονται από μια αναδυόμενη οικονομία επενδύουν δηλαδή οι επενδυτές αυτές από μια φτωχή χώρα σε μια πλούσια χώρα. Δεύτερον, ε, προσπαθούν ε, να πωλήσουν κάποια περιουσιακά στοιχεία για να είναι περισσότερο επικερδής οι επιχειρήσεις τους. Και εδώ αυτή τη φορά έχουμε το αντίστροφο φαινόμενο σε σχέση με το Μάρκο Πόλο που είχε φέρει τεχνογνωσία από την Ευρώπη στην Κίνα. Κάνουμε το αντίστροφο αυτή τη στιγμή. προέρχονται από μια χώρα που αποκαλείται κομμουνιστική και υπήρχε η οικονομία της ε, ε, η κρατική οικονομία ε, πράγμα το οποίο δημιουργούσε ένα αδιαφανές κλίμα για τις επιχειρήσεις και για την εταιρική διακυβέρνηση. Μιλάμε για ένα καπιταλισμό που καθοδηγείται από το κράτος. Το κράτος παίζει πολύ ισχυρό ρόλο στις οικονομικές επιχειρήσεις και παράλληλα η Κίνα είναι ανταγωνιστής στον τομέα της ε, ασφάλειας ε, και εδώ ε, υπάρχει το θέμα της εξαγωγής τεχνολογίας και των κινήτρων που υπάρχουν πίσω από τις επενδύσεις. Γι' αυτό βλέπουμε κάποιες ανησυχίες των επενδυτών των Ευρωπαίων επενδυτών όπως και των Ευρωπαίων πολιτικών. Αναφέρονται πολλά στα μέσα ενημέρωσης για αυτά τα θέματα και με βάση μια μελέτη που κάναμε πέρυσι, όπως είπε ήδη ο Ντάνιελ Βαντενμπούλκε, οι Κινέζοι επενδυτές δεν είναι μια ομοιογενής κατηγορία, είναι πολύ διαφορετικοί το 95% είναι ιδιώτες που επενδύουν στην Ευρώπη ή είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι κρατικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους. Οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες, μικρότερες επιχειρήσεις και υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο ως παγκόσμιοι παίκτες ε, σε κάποιες ειδικές αγορές. Μπορεί να είναι εταιρείε που στο παρελθόν παρήγαν για κάποια ε, εταιρεία, παρήγαν ε, ανταλλακτικά παραδείγματο χάρη και τώρα προσπαθούν να μετακινηθούν από το κάτω μέρος της αλυσίδας αξίας σε ανώτερο επίπεδο της αλυσίδας αξίας και τα κίνητρά τους επίσης είναι διαφορετικά. Στο παρελθόν διαβάζαμε ότι οι κινέζικες εταιρείες αναζητούσαν πόρους, αναζητούσαν τεχνολογίες, αναζητούσαν ε, εταιρικές επωνυμίες, αλλά βλέπουμε ότι πολλές εταιρείες έρχονται στην Ευρώπη επεκτείνοντας την αγορά τους, προσπαθώντας ε, να βρουν εμπορικές ε, επιχειρήσεις, εμπορικές δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν την εμπορική τους δραστηριότητα στην Κίνα. Και μερικές φορές ε, οι επιχειρήσεις τους και οι επενδύσεις στην Ευρώπη συνδέονται με το κίνητρο που έχουν ε, να μεταναστεύσουν από την Κίνα σε άλλη χώρα. Μερικές φορές ε, είναι δραστηριότητες λιγότερο γνώσεις εντατικές και χαμηλής τεχνολογίας. Ας δούμε αν ε, οι ξένες επενδύσεις από την Κίνα στην Ευρώπη είναι διαφορετικές από ότι οι ξένες επενδύσεις από την Κίνα σε άλλες χώρες. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τις κινέζικες επενδύσεις στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, βλέπουμε ότι οι, επενδύσεις, οι κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη δεν αποζητούν πόρους και δεν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν περιουσιακά στοιχεία δηλαδή δεν μεταφέρουν στην Ευρώπη την τεχνολογία τους που είναι εργασία συντατική για να παράγουν περισσότερο και αν το τη συγκρίνεται με τις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, περισσότερο αποζητούν περιουσιακά στοιχεία παρά τεχνολογία, εταιρικές επωνυμίες και αυτό διότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη ο οργανισμός που υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείε, ο CFI US, που είναι η Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες. και δεν βλέπουμε να υπάρχουν πολιτικές διενέξεις στην Ευρώπη σε σχέση με τις δραστηριότητες. Θα προσπαθήσω να καλύψω ορισμένες ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα πάρω σαν παράδειγμα τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συγχωνεύσεις. Πέρυσι ελέγχθηκαν ε, πέντε τέτοια επενδυτικά προγράμματα της Κίνας ε, για να αποδειχθεί αν υπήρχε συγκρό... Ε, συγκέντρωση βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις συγχωνεύσεις. Ένα βασικό ζήτημα είναι το πόσο μεγάλες είναι αυτές οι κινέζικες επιχειρήσεις και πού βρίσκεται το όριο μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής, κρατικής και ιδιωτικής επιχείρησης. Κάποιες επιχειρήσεις υπάρχουν ε, στον κατάλογο του Fortune Global 500 του 2011 και για τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές το βασικό αντικείμενο είναι το να καθορίσουν πόσο μεγάλες είναι οι κρατικές επιχειρήσεις. Όλες ε, οι κρατικές κινέζικες επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα φορέα ε, στην Κίνα. Και ένα σημαντικό θέμα είναι ε, ο πολιτικός έλεγχος αυτής της αρχής. Αν λοιπόν συγκεντρώσετε όλες τις κινέζικες επιχειρήσεις, θα μπορούσε κανείς να τις βάλει ε, σε μία κατηγορία και να φανεί ότι μειώνεται το μέγεθός τους εφόσον ανήκουν σε μία μόνο επιχείρηση. Και σε μερικές περιπτώσεις είναι εύκολο ε, να αποφανθούμε ότι υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές λοιπόν κατέριψαν ορισμένες υποθέσεις αλλά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτηματικά για τις κινέζικες κρατικές επιχειρήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε μία στάση αναμονής που ενδέχεται να είναι μια ορολογιακή βόμβα, γιατί αργότερα θα φανούν τα αποτελέσματά της. Θα πάρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα, θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. για κινέζικες εταιρείες που θέλουν να είναι σε θέση να μπορούν να αναδιαπραγματευτούν κάποιες συμβάσεις. Αυτό δεν ήταν εφικτό στην Ασία στην Αφρική σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αυτό είχε σχέση με την Κόβεκ στην Πολωνία που δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει τα προβλήματα. Το επόμενο παράδειγμα, η επόμενη υπόθεση είναι η Volvo όπου είχαμε το φαινόμενο της ενοποίησης της εταιρείας μετά την εξαγορά. Είναι διαφορετική αυτή η περίπτωση από ότι οι αμερικανικές εξαγορές που αμέσως μετά την εξαγορά υπάρχει μια ισχυρή ομάδα διοίκησης. Οι κινέζικες εταιρείες αποδεικνύονται ακόμη αδύναμες στην διεθνή ε, διαχείριση επιχειρήσεων, στη διεθνή διοίκηση επιχειρήσεων. Εδώ δεν έχουμε μια ορολογιακή βόμβα όπως έλεγα πριν, αλλά είναι μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν και οι τοπικές εταιρείες και οι κινέζικες εταιρείες, γιατί θα υπάρχουν ε, κενά στην τεχνολογία, θα υπάρχει μεγάλη πολιτιστική διαφορά και θα είναι πολλά τα προβλήματα για την τοπική απασχόληση. Αναβάλλεται λοιπόν η επίλυση των προβλημάτων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει οι κυβερνήσεις να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πρόκληση. Η τέταρτη υπόθεση που θα ήθελα να αναφέρω είναι η υπόθεση του Πράτο. Ξέρουμε ότι στο Πράτο είναι το κέντρο της κλωστοβιομηχανίας για την Ευρώπη. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 όμως άρχισε μία παρακμή λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών σε αυτή την περιοχή της ε, Τρίτης Ιταλίας όπως ονομαζόταν και ξέρουμε ότι οι Κινέζοι είναι πολύ ισχυροί στον ε, τομέα, έχουν πολλές ε, μεταποιητικές επιχειρήσεις με νέο μοντέλο για τις τοπικές επιχειρήσεις είναι πολύ ευέλικτες και μπορούν να παραδίδουν τα προϊόντα τους ταχύτατα σε ανταγωνιστικές τιμές και αυτό ανάγκασε ε, την περιοχή του Πράτο στην Ιταλία να περάσει από την κλωστοϊφαντουργία στον τομέα της μόδας για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους Κινέζους κλωστοϊφαντουργούς. Αυτά είναι τα παραδείγματα που ήθελα να σας αναφέρω και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η βιομηχανική αναδιάρθρωση θα είναι ένα βασικό σημείο και η εταιρική αναδιάρθρωση επίσης, όπως επίσης και οι εθνικές κοινότητες που θα πρέπει να αφομοιωθούν ή να αντιμετωπίσουν διακριτική μεταχείριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε ε, Σε μια εξαγορά επιχειρήσεων ε, είχαμε και εξαγορά Βρετανικής εταιρείας που παράγει ταξί. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντέρκ Μόνς από το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά παρακαλώ. Ελπίζω να τα καταφέρω. 14 είναι οι διαφάνειες. Uh, Έχοντα εξετάσει τις ε, κινέζικες επενδύσεις ε, στην Ευρώπη, εγώ θα έχω το προνόμιο να μιλήσω για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Κίνα, τις προκλήσεις και τις ε, δυνατότητες που, που δίνουν αυτές. Πρώτα απ' όλα η Κίνα δεν ε, έχει όλο και λιγότερη σημασία, δεν μειώνει τη σημασία της ε, 600 ε, εταιρείε απάντησαν από τις 1500 και είδαμε ότι είναι ε, ολοένα και αυξανόμενη σημασία της Κίνας για τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Για προφανείς λόγους είναι μεγάλη αγορά, εξελίσσεται ραγδαία και ένα μεγάλο τμήμα, μια μεγάλη αναλογία του παγκοσμίου εισοδήματος ε, των εταιριών προέρχονται από την Κίνα. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυξάνεται η σημασία της και δεν υπάρχει δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε είναι πρόθυμες να επενδύσουν εκεί. 63% των εταιρεών μα είπαν ότι έχουν σκοπό να κάνουν νέε επενδύσει στην Κίνα. Ε, όχι μόνο ε, άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και ε, σε εκπαίδευση, σε κατάρτιση προσωπικού, αλλά και σε κεφαλαιοχικά αγαθά. 71% από τις 600, υπηρεσί, 600 εταιρείε μας είπαν ότι η Κίνα είναι μία από τις, ένας από τους τρεις βασικούς ε, προορισμούς. Είναι πολύ σημαντική για στρατηγικούς λόγους η Κίνα και οι ευρωπαϊκές εταιρείε προτίθενται να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους εκεί. Αυτά είναι τα καλά νέα. Για γιατί δεν υπάρχουν άλλες επενδύσεις περισσότερες, γιατί υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια. Όταν τους ρωτάμε πώς βλέπετε την κυβερνητική πολιτική να επηρεάζει την καθημερινή σας δουλειά, 42% μας είπαν ότι κατά τα τελευταία δύο χρόνια δεν ε, ε, έγιναν ευκολότερα τα πράγματα. Το 42% μας είπαν ότι το περιβάλλον είναι πιο, ε, έχει περισσότερες διακρίσεις ε, ε, και αυτό είναι ένα αρκετά ανησυχητικό ποσοστό κατά τη γνώμη μου. Και βέβαια αυτό σημαίνει χαμένες ευκαιρίες, γιατί 48% μας είπαν ότι αυτό επηρεάζει το, το, το, το εισόδημά τους. Όταν τους ρωτήσαμε έχετε σκοπό να μεταφέρετε τις επενδύσεις από την Κίνα σε άλλες ε, περιφέρειες, 22% είπαν ναι. Ε, λόγω του ότι αυξάνεται το κόστος ε, το μισθολογικό αλλά και το, το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι διαφορετικό και βέβαια επίσης η σχετική ελκυστικότητα άλλων ε, περιφερειών είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος η αλλά υπάρχουν και άλλες αγορές και οι εταιρείε προφανώς προσπαθούν να δουν να, να υπάρχει μια ισορροπία. οι κρατικές ε, επιχειρήσεις, ε, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που έχουν συμφέροντος στο εξωτερικό τυχαίνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Συχνά υπάρχουν μονοπόλια, διοικητικά, υπάρχουν ρυθμιστικά πλεονεκτήματα για τις κρατικές επιχειρήσεις, ε, καλύτερη πρόσβαση σε φθηνούς πόρους, ενώ οι ιδιωτικέ κινεζικέ επιχειρήσεις έχουν σημαντικές δυσκολίες και το ίδιο ισχύει και για τις ε, επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων. Ε, ε, επομένως οι εταιρείες αυτές έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα, παροχημένα συστήματα διοθότησης, υποχρέωση κοινοπραξίας, να μπει κανείς σε μια κοινοπραξία για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στην αγορά και βεβαίως σε μεγάλο βαθμό αποκλείονται από τη διατύπωση των προτύπων που de facto μπορεί να είναι μη δασμολογικό εμπόδιο για την ε, ε, είσοδο στην κινέζικη αγορά. Στο πρόσφατο έγγραφο θέσεώς μας που ετησίως δημοσιεύουμε αναγνωρίσαμε όχι μόνο εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά αλλά και πέντε είδους, είδη συμπεριφοράς που θεωρούμε ότι πρέπει να ε, εξεταστούν γιατί είναι πηγή ανισότητας. Δηλαδή πρόσβαση στην αγορά, ε, υπάρχει το θέμα και επίσης των δημόσιων προμηθειών. Είναι μια τεράστια ευκαιρία πιστεύουμε για τις ευρωπαϊκές ε, εταιρείε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο τομέα να έχει κανεί πρόσβαση δηλαδή στον τομέα αυτό. Υπάρχει και θέμα ε, του πώς μεταχειρίζονται οι Κινέζοι τις διάφορες εταιρείες σε επίπεδο ε, νομοθεσίας, το θέμα του κράτους δικαίου δηλαδή, το κράτος δικαίου και επίσης ε, αναφέρθηκα και στα ζητήματα των τεχνολογιών ε, και των υπηρεσιών. Πιστεύουμε λοιπόν ως προς την πρόσβαση στην αγορά ότι υπάρχουν πέντε τομείς όπου υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, υπάρχουν πλήρως προστατευμένοι τομείς ε, οι οποίοι είχαν νόημα πριν από 10 χρόνια όταν μπήκε πρώτη φορά στον ΠΟΕ εκείνα αλλά άλλαξαν τα πράγματα και τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και βλέπουμε σε αυτούς τους τομείς που τώρα φεύγουν από την Κίνα και δραστηριοποιούνται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο οπότε πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί όλο, όλο αυτό το θέμα των πολιτικών των πλήρως προστατευμένων ανέφερα το θέμα της απέτηση κοινοπραξίας ε, που είναι ένας τρόπος μεταφοράς τεχνολογίας γιατί αν θέλει κανείς να μπει στην αγορά χρειάζεται κοινοπραξία και ο εταίρο θα σου ζητήσει να, σου, να μεταφέρεις κάποια ε, τεχνογνωσία, διαφορετικά δεν υπάρχει κοινοπραξία ούτε πρόσβαση στην αγορά. Ε, οι απαιτήσει για την αδειοδότηση επίσης είναι ένας τομέας που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να διευκολυνθούν κάπως τα πράγματα. Είναι διαφορετική η μεταχείριση. Οι κινέζικες εταιρείε ε, όταν ζητούν δηλαδή μια άδεια είναι διαφορετική διαδικασία και διαφορετική για τι υπόλοιπε εταιρείε. Αξιώσεις για την εθνική ασφάλεια. Δεν είναι πολύ σαφέ τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ε, είναι πάντως ένα μη δασμολογικό εμπόδιο όπω τα προηγούμενα που ανέφερα. Θα τα πω γρήγορα, οι διμερείς επενδύσεις ε, είναι ακόμη σε χαμηλό επίπεδο για την ώρα, σε είναι δηλαδή 3,5% από την Κίνα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 2% αλλά αυξάνονται τα ποσοστά αυτά. Ο συνάδελφος Φαντεμπούκε το είπε άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον το εμπορικό επιμελητήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα ε, υποστηρίζεται, θεωρούμε ότι είναι κάτι το καλό ε, ότι ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, ότι πιέζει τις ε, εγχώριε εταιρείε, θεωρούμε ότι είναι κάτι το καλό. Υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη η Κίνα να σκεφτεί και να εξετάσει το, το εξή γεγονό, ότι όλο και περισσότερε επενδύσει υπάρχουν από την Κίνα στην Ευρώπη, σε τομεί όπου οι ευρωπαϊκέ ε, εταιρείε δεν μπορούν στην Κίνα να έχουν πρόσβαση. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ του τι κάνουν οι κινεζικέ εταιρείε στην Ευρώπη και ε, μεταξύ του τι κάνουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε στην Κίνα. Αυτό το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί προς το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά και προς όφελος της Κίνας, γιατί αν δεν καλυφθεί αυτό το, το χάσμα, θα υπάρξει πλέον αντίσταση στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτή η αντίσταση μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες επενδύσεις και λιγότερες ευκαιρίες ε, επενδύσεων για την Κίνα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη συνθήκη ή συμφωνία. Πιστεύω ότι μία ενδεχόμενη συνθήκη θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις επενδυτικές πραγματικότητες που μόλις ανέφερα, όχι δηλαδή ε, μόνο το θέμα της εθνικής ε, μεταχείρισης μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης, αλλά και πριν από την ε, εγκατάσταση της επιχείρησης, για τους λόγους που μόλις ανέφερα. Τι λοιπόν θα μπορούσε συγκεκριμένα να γίνει ως προς αυτό, ε, τα εμπόδια που ανέφερα ε, για το έγγραφο που καλύπτει 45 κλάδους, 45 συστάσεις πολύ συγκεκριμένες για την πρόσβαση στην αγορά, ενδεχομένως αυτό είναι κάτι που πρέπει να ε, το δούμε. Ε, όσον αφορά τώρα τον κατάλογο ξένων επενδύσεων, πιστεύουμε ότι αυτός, αυτό είναι ένα εργαλείο λίγο αναχρονιστικό, αλλά στην αρχή όταν αναπτυσσόταν η Κίνα ήταν χρήσιμο. Σήμερα όμως ε, οι περισσότεροι από τους τομείς αυτός ε, ε, που επιτρέπονται αλλά και που απαγορεύονται, πρέπει να ανοίξουν περισσότερο προς τα έξω και υπάρχουν και κάποιοι τομείς όπου υπάρχουν διοικητικά μονοπόλια και πιστεύω ότι επιτέλους έχει έρθει η ώρα να ανοίξουν οι τομείς αυτοί και αυτό είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει και η κινέζικη κυβέρνηση. Υπάρχει επίσης, υπάρχουν και οι κλασικοί ε, όροι προστασίας των επενδύσεων, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Thank you, Mr. I was... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ με ενδιαφέρει αυτό που είπατε για τις επενδύσεις στην Κίνα και την πρόσβαση στην αγορά. Είναι πραγματικά ζητήματα για τα οποία συμφωνώ απολύτως. Ε, είναι ενδιαφέρον πιστεύω για μας ε, να ακούσουμε εκείνους που είναι πράγματι εμπλεκόμενοι φορείς που όντως ε, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κίνα. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε ερωτήσεις, ελπίζω και απαντήσεις, να δώσω το λόγο στον Χέλμου Τσόλς που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας για την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, από την πρώτη ενότητα γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Πρέπει να βρούμε ε, τη σωστή οπτική γωνία για να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Οι εισαγωγικέ ομιλίες έδειξαν ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα του πώς θα χειριστούμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Κίνα και αντιστρόφως τις κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη. Εξέτασα κάποια σχετικά κείμενα για να προετοιμάσω ε, τη σημερινή ακρόαση και ε, βρήκα ένα κείμενο του Henry Kissinger που ίσως να το είχατε διαβάσει όταν το είχε γράψει. Περιγράφει την ε, επίσκεψή του στην Κίνα το 1973 και σκεφτόταν πώς να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις πώς να βρεθεί μια κοινή, ένα κοινό πεδίο συνεννόησης για να επιληθούν τα προβλήματα. Βέβαια το 1973 δεν ήταν η κατάσταση ίδια με σήμερα. Και ε, γράφει ότι δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς ε, ήδη έχοντας ένα συμβιβασμό στο μυαλό του. Πρέπει να βάζει ε, κανείς ε, σε ίση θέση τις απόψεις των δύο πλευρών και να, από αυτό να προκύπτουν τα βασικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Και νομίζω ότι και για την Ευρώπη η πρόκληση σήμερα είναι το να βάλουμε επιτάπητο σε αυτά τα οποία θέλουμε από την κινέζικη αγορά, ποια είναι τα συμφέροντά μας και να καταλάβουμε και ποια είναι τα συμφέροντα της κινέζικης οικονομίας και των Κινέζων που έρχονται στην Ευρώπη και να δούμε κατά πόσο μας συμφέρει και εμάς να έρχονται Κινέζοι επενδυτές στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου είναι ένα τμήμα μόνο της ε, Ευρώπης. Και μας υπενθύμισε ο καθηγητής στην ομιλία του ότι και η Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι τμήμα της Ευρώπης και επενδύουν και εκεί οι Κινέζοι. Η σημερινή ακρόαση θα πρέπει να συνεισφέρει ακριβώς σε αυτή την κατανόηση. Δηλαδή ότι όταν μιλάμε για ε, τις επενδυτικές πολιτικές των δύο οικονομικών εταίρων θα πρέπει να θεσπίσουμε αξιόπιστη νομοθεσία που θα βοηθήσουν τους επενδυτές να συνεισφέρουν ε, στην ισχυροποίηση και των δύο οικονομιών. και το πρωί που συζητούσαμε τα όσα ανέφερε η ομάδα παρακολούθησης της Επιτροπής μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Κίνα 1,3 δισεκατομμύρια πολίτες που καταναλώνουν όπως καταναλώνουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Κινέζοι πρέπει να αναζητήσουν πρώτες ύλες κάπου. Χρειάζεται λοιπόν μια ανοιχτόμυαλη πολιτική για, τους, ε, για τις πρώτες ύλες και για τους πόρους που αναζητούν στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού, όπως και εμείς στην Ευρώπη αναζητούμε πόρους για την παραγωγή μας. Θέλουμε και οι δύο οικονομικοί εταίροι να μπορέσουν να συνεισφέρουν ε, στην ενίσχυση και στην αναδιοργάνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι νομίζω πρέπει να κρίνουμε τα κριτήρια για την επενδυτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κίνα. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω εισαγωγικά. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία μελέτη για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και εκφράζονται αρκετές ανησυχίες για τις κινέζικες επενδύσεις. Οι ανησυχίες αφορούν ε, ε, τις πολιτιστικές διαφορές, το ότι η Κίνα αγνοεί πολιτικές και νομοθεσίες ε, που έχουν σχέση με ε, την ε, μείωση του διεξιδίου του άνθρακος και την βιωσιμότητα. Οι Κινέζοι επενδύουν ε, εστιάζοντας στο βραχυπρόθεσμο όφελος. Δεν υπάρχει διαφάνεια στην Κίνα. Έλλειψη κατανόησης και αυταρχικός χαρακτήρας του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Αναφέρω αυτά τα στοιχεία από αυτή τη μελέτη γιατί δίνει κάποια παραδείγματα για το φόβο της ευρωπαϊκής οικονομίας για τις κινέζικες επενδύσεις. Και αυτό είναι μία από τις προκλήσεις. Πρέπει να σας πω εξ ότι εγώ δεν συμφωνώ με τα απορίσματα αυτής της μελέτης. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μία άλλη προσέγγιση. Στη Γερμανία ένα ντοκιμαντέρ την περασμένη εβδομάδα έδειξε πώς άλλαξε η ιδιοκτησία μιας επιχείρησης ε, και οι υπάλληλοι μιας εταιρείας καθαρισμού ε, χαίρονται που πέρασε η ιδιοκτησία σε Κινέζους διότι διατηρούν τις θέσεις απασχόλησής τους και παράλληλα μπορούν και να ε, υπερασπίσουν ε, τα εργατικά τους δικαιώματα. Ε, γνωρίζουμε επίσης και το παράδειγμα της Κόσκο στον Πειραιά όπου η κινέζικη ιδιοκτησία θέτει σε κίνδυνο τα εργασιακά δικαιώματα των Ελλήνων που απασχολούνται εκεί ή των ε, εργαζομένων από άλλες χώρες στην Ελλάδα. Δημιουργείται δηλαδή ένα είδος ανταγωνισμού μέσα στο εργατικό δυναμικό. Και αυτό θέτει το ερώτημα του αν συνδέουμε τις επενδυτικές πολιτικές που μόλις αρχίσαμε να συζητάμε με κριτήρια οικολογίας, ε, εργασιακών δικαιωμάτων που θα πρέπει ισότιμα να τεθούν για τις κινέζικες ή ευρωπαϊκές επενδύσεις στην αντίστοιχη χώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτσο και κυρία Ντεσσαρνέζ. Ναι, ευχαριστώ. Δύο θέματα για τις επενδύσεις. Μόλις το είπε και ο Σναφος Σόλτς. Πρώτα απ' όλα θέμα διαφάνειας δεν είναι πολύ σημαντικέ οι επενδύσει κινέζικε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλη την ε, αύξησή του με σταθερομαριθμό. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε την εγγνευσιμότητα από πού έρχονται, τι είναι στρατηγική σημασία, ε, εξαγορέ επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη στήριξη, είτε για να του πάρουν ε, τι διάφορε άδειε εκμετάλλευση και να τι αφήσουν είτε στρατηγικές που έχουν να κάνουν με ναυτιλιακή μεταφορά το ένα το άλλο. Και όπως στις ΗΠΑ υπάρχει μια διαφάνεια για τις ε, επενδύσεις απ' έξω, το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κινέζικες επενδύσεις. Και εδώ ένα μισή χρόνο αναρωτιόμαστε τι γίνεται με τις στην Ευρώπη επενδύσεις της Κίνας και όταν έθεσα το ερώτημα για την αριθμότητα αυτών δεν μου έδωσε καμιά απάντηση. Ναι, αλλά έχουν ε, σημειωθεί αυτές οι επενδύσεις και κρίμα είναι και ίσως ε, ευνοούν και διάφορες αμφιβολίες και υποψίες που δεν χρειάζονται και ακόμα για τις επενδύσεις της ευρωπαϊκές ξένες στην Κίνα. Εκεί τίθεται το ερώτημα και στο σύνολο της διαδικασίας του joint venture είναι μια μεταφορά σχεδόν αυτόματη τεχνολογίας για να μπορέσει κανείς να προσεγγράψει ένα συμβόλαιο με Κινέζους εταίρους. Και αυτό δημιουργεί ένα κάποιο πρόβλημα από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε και με κοινοπραξίες ακριβώς και στην Κίνα. Η μεταφορά τεχνολογίας αυτό δημιουργεί πρόβλημα και νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα για όλους τους Ευρωπαίους. Τρίτο θέμα που θέτω επιτάπητος είναι η αρχή της αμοιβαιότητας. Εντάξει, τα πάντα μπορούν να ισχύουν από τη στιγμή όμως που υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Ορισμένε ε, δημοσιαγορέ να ανοίξουν σε επενδύσει, αλλά υπάρχει η απαραίτητη αντιστοιχία και στην Κίνα. Αυτό ήθελα να πω τώρα σε αυτή τη φάση τη συζήτηση και ευχαριστώ ιδιαίτερα του συναδέλφους που οργάνωσαν το hearing αυτό ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Ναι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ επίκαιρη η ακρόασή μας γιατί την περασμένη εβδομάδα εμείς στην αντιπροσωπεία των σχέσεων με την Κίνα πήγαμε στην Κίνα και γνωρίσαμε το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, ήταν λίγο διαφορετική η ατμόσφαιρα από τη σημερινή εδώ. Έχω ε, μία παρατηρήση. Όταν μιλάμε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας οι δημόσιες δηλώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, ε, περιεκτική ε, συνεργασία, ε, στρατηγική συνεργασία με την Κίνα. Όταν όμως περνάμε στην πράξη βλέπουμε 4, 5, 6 διμερείς δεσμεύσεις και κάποιες ε, λιγότερο σημαντικές δεσμεύσεις ε, επιπλέον σε ένα πολύ μεγάλο πακέτο το οποίο είναι κάπως αόριστο. Δεν φταίει η Κίνα, εδώ φταίει η Ευρώπη. Οι συνομιλητές μας στο Πεκίνο αλλά και στην Ευρώπη πιστεύουν ότι η βασική μας αδυναμία σε οποιαδήποτε μας σχέση με την Κίνα είναι η ικανότητά μας ε, να καθορίσουμε μία αποτελεσματική στρατηγική με την Κίνα και πώς μπορούμε να συγκεράσουμε πολύ ισχυρές διμερείς δεσμεύσεις που προέρχονται κυρίως από τις μεγαλύτερες χώρες, από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες στρέφονται προς την Κίνα και θεωρούν ότι είναι προνομιούχος συνομιλητής τους. Δεύτερον, όταν μιλούμε για συμμετρικές ε, και τέλος πάντων παρόμοια μεταχείριση για τις κινέζικες και ευρωπαϊκές εταιρείες. Στη Μόφκομ έγινε μία συζήτηση, συνάντηση και ένας εξέχων συνάδελφος του ΕΛΚ είπε το εξής. Γιατί δεν υπάρχει συμμετρική μεταχείριση των δύο ε, μερών και οι, κινέζικες, ε, οι, Κινέζοι μας, οι συνομιλητές μας μας απάντησαν Μα θέλετε να έχουμε συμμετρική μεταχείριση στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ε, γιατί η οι δικέ σας εταιρείε θα ελέγχουν τη δική μας αγορά πάνω από 50% και εμεί θα ελέγχουμε τόσο λιγότερο τις δικές σας, ε, τη δική σας αγορά στην ε, Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψη στρατηγικής τη Ευρώπη ενώπιον της Κίνα και θα ήταν πραγματικά ένα ακαδημαϊκό εγχείρημα αυτό που θα έπρεπε να γίνει ενδεχομένω πρέπει να συζητήσουμε με την Κίνα ως Ευρώπη και όχι μόνο ως Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία και ούτω καθεξής. Όσο συζητούμε διμερώς εκ μέρους των κρατών μελών μας, χάνουμε το ανταγωνι... τον ανταγωνισμό μας, ε, ε, τον... χάνουμε στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Και επίσης αν ε, η επενδυτική μας συμφωνία δεν είναι περιεκτική και δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα 27 κράτη-μέλη, πάλι ένα χαρτί θα είναι μόνο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους τρεις προσκεκλημένους μας στο πάνελ να απαντήσουν uh, πολύ σύντομα σε αυτά που άκουσαν. Όσο το δυνατόν συντομότερα παρακαλώ. Θα σχολιάσω πολύ σύντομα μετά από αυτά τα οποία μόλις είπε η κυρία Ντεσαγνέ. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το, το θέμα των σχέσεων και είπε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θα πρέπει να προσπαθήσουν να μας δώσουν περισσότερα δεδομένα για αυτές τις επενδύσεις. Και ένα θέμα που επίσης ανέφερα είναι ότι δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα πολύ καλά την πολιτική καινοτομία της Κίνας και το κατά πόσο λειτουργεί αυτή η πολιτική και το θέμα της αμοιβαιότητας. είναι σημαντικό και θα είναι ένα από τα δύσκολα θέματα. Και ελπίζω ότι οι ευρωπαίοι, οι πολιτικοί θα μπορέσουν να το χειρίσουν αυτό το θέμα. Θα μιλήσω και για αυτό το τελευταίο θέμα για την ε, πολιτική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κίνας. Έχουμε δει ότι τα κράτη-μέλη ακολουθούν διαφορετική στάση όσον αφορά την καταγραφή ε, των επενδύσεων. Ο ΣΑ δημοσιεύει ένα κατάλογο και ορισμένε χώρε ε, είναι πολύ ανοιχτέ στο στάδιο των ρυθμίσεων πριν από την εγκατάσταση. Άλλε χώρε είναι αυστηρέ κατά την επιχειρησιακή φάση, δηλαδή μετά την εγκατάσταση. Και αν ε, τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, φαίνεται ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή πολιτική άμεσων ξένων επενδύσεων για να συντονίζει την πολιτική των κρατών μελών ανεξαρτήτως μεγέθους. Ευχαριστώ. Um, να προσθέσω κάτι σε αυτά που μόλις είπαν οι δύο συνάδελφοι για τη μεταφορά τεχνολογίας. Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι, ότι η μεταφορά τεχνολογίας είναι μια επιχειρηματική απόφαση και όχι ένα τίμημα για να έχει κανείς πρόσβαση στην αγορά και αυτό είναι ένας από τους τομείς τους οποίους έχουμε εντοπίσει όπου δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση και εδώ θα πρέπει να υπάρξει. Και είναι προς όφελος της Κίνας, προς συμφέρον της Κίνας το να γίνει αυτό γιατί Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη προστασία των, της τεχνολογίας από τη στιγμή που μεταφέρεται και γι' αυτό οι εταιρείε δεν δίνουν την τεχνολογία εχμής. Αλλά αν δεν δώσουν την τεχνολογία εχμής δεν συνεισφέρουν στην ε, οικονομία της Κίνας. Και νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε θα μπορούσαν να συνεισφέρουν καλύτερα και περισσότερο εάν οι αποφάσεις βασίζονται σε επιχειρηματικά κριτήρια για την μεταφορά τεχνολογίας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο για την αμοιβαιότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία κατά τη γνώμη μου ότι η Ευρώπη είναι πιο ανοιχτή από την Κίνα. Και ευχαρίστω ε, οι συνάδελφοι από την Μόφκομ να έρθουν να το συζητήσουμε, να ακούσουμε τι έχουν να πούν για το έγγραφο το οποίο δέκα χρόνια τώρα ε, ε, εκδίδουμε. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει και να παραμείνει ανοιχτή η Ευρώπη. Όταν μιλάμε για αμοιβαιότητα, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για επικοδομητική και θετική αμοιβαιότητα. Να καταβάλουμε προσπάθειες να εξηγήσουμε στην Κίνα ότι είναι προς συμφέρον της να εξετάσει την ε, κατάσταση στην Κίνα, διότι αν δεν το κάνει αυτή η πολιτική αντίσταση ε, θα φτάσει και στην ευρωπαϊκή ε, αγορά, θα δυσκολεύσει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Θέλουμε λοιπόν να πείσουμε την Κίνα να ακολουθήσει μια θετική πορεία, ότι δηλαδή η πιο ανοιχτή στάση της Κίνας είναι καλύτερη λύση και όχι το κλείσιμο της ευρωπαϊκής αγοράς. Ευχαριστώ. Εποφελούμενος της ευκαιρίας, θα ευχαριστήσω τους τρεις διακεκριμένους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους, γιατί ήταν μια συζήτηση αποκαλυπτική και πολύ χρήσιμη για όλους μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρουσίαση των θέσεών σας. Ο Χέλμουτ είναι ο εισηγητής μας, ο μόνιμος εισηγητής για την Κίνα και εγώ είμαι μέλος της μόνιμης ομάδας αυτής. Και θέλω να πω ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπατε. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και πολύ κίνδυνοι παράλληλα στις επιχειρήσεις πάντοτε υπάρχει και ο κίνδυνος όταν επιζητούμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Ήταν μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα θα δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε τώρα ή θέλετε να μιλήσετε στο τέλος. Στον κύριο Wen Huashan από την Κίνα και αν και κάποιος εκπρόσωπος της Επιτροπής να λάβει το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε τώρα ή στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερως που βρίσκομαι σήμερα εδώ. και θα ήθελα να μην με τρόμαζαν οι παρατηρήσεις που άκουσα μέχρι τώρα. Συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Γιατί οι κινέζικες επενδύσεις ε, προτιμούν την Ευρώπη από ότι άλλα μέρη του κόσμου. Η απάντηση είναι ότι δεν, υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχουν πολιτικές διενέξει και μπορούμε να έχουμε καλύτερο επενδυτικό κλίμα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την Κίνα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές επενδύσεις στην Κίνα. Ε, θέλω καταρχήν να μιλήσω για τις κινέζικες επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής Τσάνγκ στην ε, υπόθεση που αφορούσε τη Βόλβο, Ένα πλεονέκτημα για τις κινέζικες επενδύσεις, τις επενδύσεις ε, από μεγάλες εταιρείες κυρίως, είναι ότι στη διαδικασία αυτή ε, συνεχώς ε, διδάσκονται και θα πρέπει να σέβονται τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις. Ε, ε, επισκέφθηκα το ε, μεγαλύτερο εργοστάσιο της Volvo στη Γκέντ και μου έκανε εντύπωση μία επιγραφή που διάβασα που έλεγε η Volvo είναι Volvo και η Geely είναι Geely. Τα τελευταία δύο χρόνια η Volvo έχει αυξήσει την παραγωγή της και ένας λόγος είναι ότι ε, υπάρχει ροή κεφαλαίου από την Τζίλη και αυτές οι επενδύσεις έχουν δημιουργήσει μια ευρεία αγορά για τις τοπικές εταιρείες. Ένα τρίτο σημείο. Όσον αφορά το τοπικό επίπεδο. Το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι που μίλησαν και για την μεταφορά τεχνολογίας. Η Κίνα έχει συμφωνήσει να δεχθεί τα πρότυπα ΑΠΕΚ και θα δείτε ότι όλες οι διεθνείς επενδύσεις, είτε συμφωνίες ε, ελεύθερου εμπορίου, είτε διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, δεν αναφέρουν το τοπικό επίπεδο. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν για τη μεταφορά τεχνολογίας από όσο θυμάμαι στις μεταφορές τεχνολογίας δεν ε, μιλάμε για απαιτήσει από κρατικής πλευράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι επιχειρηματική συμπεριφορά, όπως και οι Κινέζοι να ζητούν Ευρωπαίους εταίρους για να κάνουν μια κοινοπραξία. Ή θα βάλεις χρήματα ή θα βάλεις κάτι άλλο. Αν δεν έχεις χρήματα, κάτι πρέπει να βάλεις. Είναι μια απλή φιλοσοφία. Δύο επιχειρηματικοί εταίροι για να κάνουν μια κοινοπραξία πρέπει και οι δύο να συνεισφέρουν. Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σας για τη μεταφορά τεχνολογίας. και η αγαπητή ε, κυρία από τη Γαλλία ε, μας είπε κάτι το οποίο όντως ε, γνωρίζω. Όταν μιλάμε για κινέζικες επενδύσεις, συχνά θέλουμε να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα χρήματα. Ο Υπουργός Οικονομίας της Κίνας κατέληξε σε συνένεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι και οι δύο πλευρές θα δεχθούν αυτή την ε, λογιστική εγγραφή εάν τα χρήματα δεν είναι παράνομα είναι θέμα λογιστικής το να βρεθεί από πού προέρχονται τα χρήματα. Και έχουμε φτάσει σε συνένεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της προέλευσης των χρημάτων. Άρα νομίζω ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις του από πού προέρχονται τα χρήματα ελπίζω ότι στο μέλλον δεν θα αποτελούν πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λεοπόλ Ρουμπινάκη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, ε, παρουσιάσεις αυτές που ακούσαμε από τους τρεις προκεκλημένους σε αυτό το πάνελ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Όπως ε, γνωρίζετε ε, στη συνέχεια των εξελίξεων που, που αναφέρατε στην, στα εισαγωγικά σας σχόλια, δηλαδή τη σύνοδο, την επιχειμένη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ε, για την επενδυτική συμφωνία, θα γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει συμπεριλάβει ε, ιδιαίτερη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και η διαβούλευση αυτή ε, συμφωνεί με πολλά από αυτά που είπαν οι προσκεκλημένοι. Η Κίνα είναι ένας πολύ σημαντικός προορισμός για τις ξένες επενδύσεις όχι, της Ευρώπης, όχι σε καθαρά νούμερα ίσως, ε, αλλά για τη στρατηγική των ευρωπαϊκών εταιριών. Και ο λόγος ε, για τον οποίο Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι η κινέζικη επένδυση είναι σημαντική ε, στην Ευρώπη. Η κινέζικη επένδυση στην Ευρώπη είναι σημαντική. Ε, είναι ισχύει και, και ισχύει εκατέρωθεν. Ε, η, Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις και στις κινέζικες. Θεωρούμε ότι είναι αρκετά κλειστή ακόμα η ευρωπαϊκή αγορά για τις κινέζικες επενδύσεις. Υπάρχουν ακόμη εμπόδια που παρακολύουν ή περιπλέκουν τις επενδύσεις ε, ε, στην Κίνα που έχουν να κάνουν με αδειοδότηση, υπάρχουν τα θέματα διακριτικής άνησης μεταχείρισης, όλα αυτά είναι ζητήματα ε, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις ενδεχομένως, τις οποίες ε, προετοιμάζουμε. δεν ε, θα είναι εύκολη ε, η διαπραγμάτευση. Περιμένω το δεύτερο πάνελ να μας εξηγήσει πώς ε, θα έχουν τα πράγματα το γεγονός ότι αυτό αποτελεί πλέον τμήμα της στρατηγικής υπό, υπό τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τη σχέση με την Κίνα πιο πολύ ως Ευρώπη και όχι ως σύνολο διμερών ε, συμφωνιών των μεμονωμένων κρατών μελών. Το θέμα των δημοσίων ε, προμηθειών βεβαίως είναι σημαντικό. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε κάπως ξεχωριστά σε σχέση με τις ε, επενδύσεις. Όσον αφορά τώρα τις στρατηγικές αναθεωρήσεις, προφανώς αυτό είναι κάτι που για την ώρα λαμβάνει χώρα σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν αυτές τις ε, αναθεωρήσεις. Το ζήτημα της ανάπτυξης ενός ε, συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είναι εκρεμές, είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα όταν κατά την εξέταση ενός, ε, μιας τέτοιας περι, πιθανότητας υπάρχουν τα θέματα της αναλογικότητας, της διαφάνειας, ε, ε, της αξιοπιστίας και της διατήρησης της δυνατότητας επενδύσεων. Το ζήτημα είναι, της, είναι βασικό το ζήτημα της διαφάνειας είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί και Επ' αυτού νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω προβληματισμός από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε το επόμενο πάνελ. Θα θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο γύρο ε, και να περάσουμε στο δεύτερο. Ε, είναι δύο ε, ακαδημαϊκοί εδώ, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν ενδεχομένως αμφιβολίες και υποψίες σε σχέση με αυτήν την επενδυτική συνθήκη πρώτη παρουσίαση Λουγ Σκόφκαρ Πούλσεν. Ο Δόκτωρ Πούλσεν ε, είναι ε, δανός ε, και αυτή τη στιγμή ερευνητής στο Νάφιλ College στην Οξφόρδη για ζητήματα επενδύσεων. Έχει δημοσιεύσει σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, πονήματα για τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες ε, που έχουν άμεση σχέση με τις αξιώσεις που βασίζονται στις διμερείς επενδυτικές συνθήκες όπως επίσης και για την διάδοση των σημερινών επενδυτικών συνθήκων και τη σημασία τους για, την, για τις εγγυήσεις ε, ε, σε σχέση με τους κινδύνους. Είναι ειδικό σε θέματα διμερών επενδυτικών συμφωνιών και σύμβουλος κρατών μελών ε, για, για, τις, για διεθνείς επενδύσεις. Ο δεύτερος προσκεκλημένος, ο καθηγητής Βένου Ασουάν, από το Τσιάντζαοτόγκ Πανεπιστήμιο της Κίνας, είναι στο Oxford Brooks University από το 2002. Ε, το 2004 ε, βρισκόταν στο ε, Cambridge. Δεν είναι μόνο ακαδημαϊκός, αλλά ασκεί το το επάγγελμα του νομικού σε επιτροπές διαιτησίας έχει ασχοληθεί κυρίως με τις ξένες επενδύσεις, ε, με τις επενδυτικές ε, πρακτικές της Κίνας και τις σχετικές συνθήκες. Ε, είναι μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Συγκριτικού Δικαίου στη Χάγη και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που άκουσα ότι πήγε στο Cambridge. Συγγνώμη, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, για το Cambridge. Να δώσω τώρα πρώτα το λόγο στον ε, δόκτωρα Πούλσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι συμμετείχα στην μελέτη που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον οικονομικό αντίκτυπο μιας ε, επενδυτικής συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, όμως εδώ είμαι ως ε, ιδιώτης και δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ότι οτιδήποτε πω είναι θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε ότι αυτά που λέω προκύπτουν από τη μελέτη αυτή, είναι στο πλαίσιο της μελέτης αυτής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους όσους βρίσκονται ε, εδώ ότι το να συμφωνήσει κανεί σε μια τέτοιου είδου συνθήκη είναι σημαντική ε, υποχρέωση για κάθε κυβέρνηση. Υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι ε, καθορίζουν ζητήματα δημοσίου δικαίου και καθορίζουν κατά πόσο είναι θεμητό να αρθούν εμπόριδια που αφορούν το περιβαλλοντικό δίκαιο, ε, για τη ρύθμιση της δημόσιας υγείας, τη φορολογία κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, προσφυγή στη συνέχεια. Είναι ένα ζήτημα, είναι, ένα, είναι μια κατάσταση πολύ μοναδική σε διεθνές επίπεδο και είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή μέσο ε, που ε, ασχολείται με την οικονομική παγκοσμιοποίηση. Θα ασχοληθώ λοιπόν σήμερα με ένα συγκεκριμένο θέμα και κατά πόσο θα έπρεπε να περιμένουμε μια επενδυτική συνθήκη Ό,τι και αν κάνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, ό,τι και αν καλύπτει, κατά πόσο θα έχει ένα πραγματικό αυτό αποτέλεσμα στις επενδυτικές ροές μεταξύ αυτών των δύο ε, ε, φορέων. Ε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι κυβερνήτες μπορεί να θέλουν να μπουν σε μια επενδυτική συνθήκη. Μπορούμε να σκεφτούμε πολλούς λόγους για τους οποίους οι επενδυτικές συνθήκες είναι χρήσιμες στους πολιτικούς. Ε, μπορώ να πω γιατί πολλέ, είναι πολύ χρήσιμες για τους γραφειοκράτες αυτές οι συνθήκες. Αλλά ένας βασικός λόγος, αν όχι ο πιο βασικός, για τον οποίο αναλαμβάνουν για χρόνια οι υποχρεώσει ε, τις υποχρεώσεις αυτές οι κυβερνήσεις είναι η πεποίθηση ότι θα έχουν αποτέλεσμα στην προθυμία των ξένων επενδυτών να επενδύσουν κεφάλαιο στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι άμεσο ή έμεσο αυτό το κεφάλαιο, σίγουρα ε, αυτό το, αυτός ο αντίκτυπος, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένας αντίκτυπος. Για μένα αυτό σημαίνει ότι το απλό γεγονός ότι μια επενδυτική συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ε, θα μπορούσε να αρχίσει να ισχύει, θα προωθούσε μεγαλύτερη συνοχή και ε, περισσότερες επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των δύο ε, φορέων. Αυτό όμως δεν είναι επαρκές επιχείρημα από μόνο του για την ε, έναρξη διαπραγματεύσεων, ούτε είναι επαρκές επιχείρημα για διαπραγματεύσεις που, που το γεγονός ότι η επενδυτική αυτή συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα διαιτησίας που στο παρελθόν δεν ίσχυε. Δεν μπορεί να είναι στόχος πολιτικής από μόνος του μπορεί όμως να είναι ένας τρόπος να επιτύχουμε ένα σκοπό και μπορεί αυτό να αυξάνει την εθνική ευημερία και ε, στις δύο περιπτώσεις. Εγώ λοιπόν βασίζομαι στην υπόθεση και μπορεί να είναι λάθος αυτό ότι οι επενδυτικές ε, ε, συνθήκες έχουν σημασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κίνα. Ε, το βασικό λοιπόν στοιχείο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι κατά πόσο αναμένεται να έχει αυτό αποτέλεσμα στην ύπαρξη ξένων επενδύσεων. Αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό επιχείρημα για την έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά αν δεν είναι, τότε χρειαζόμαστε άλλα πολύ ισχυρά επιχειρήματα για να αρχίσουμε μία δαπανηρή και μακρόχρονη διαδικασία διαπραγματεύσεων ε, ε, και υποχρεώσεων και για, τις, ε, και για τους δύο φορούς. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες στατιστικών δεδομένων γιατί δεν ε, υπάρχουν ε, ε, αρκετά στοιχεία και δεν μπορούν να είναι υψηλού επίπεδου οι αξιολογήσεις τουλάχιστον για σοβαρές οικονομίες. Είναι πιο σημαντικό να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι ίδιοι επενδυτές. Έχουμε πολλές έρευνες από τα τελευταία χρόνια, μερικές καλύπτουν και την Κίνα. Οι περισσότερες από αυτές έχουν περιορισμένη αξία γιατί έχουν ε, είναι, είναι κακή ε, η διατύπωση των ερωτήσεων, η εκφώνηση των ερωτήσεων. Οι επενδύσει δεν θα πούνε ποτέ βεβαίω ότι δεν του αρέσει μια επενδυτική συνθήκη, θα θέλουν πάντοτε ένα επιπλέον ε, επίπεδο προστασίας, άρα το βασικό ερώτημα για τους υπεύθυνου λήψη αποφάσεων και εδώ σε αυτή την αίθουσα δεν είναι κατά πόσο ε, οι επενδυτές θα ήθελαν μια τέτοια συνθήκη, αλλά αν θα έπαιζε ε, ρόλο στις επενδυτικές αποφάσει και κατά ποιο τρόπο. Το 2000, ε, το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία έρευνα 300 επενδυτών σε σχέση με, την, με τη στάση τους απέναντι σε αυτές τις επενδυτικές ε, συνθήκες και ειδικότερα τις διμερείς και η ερώτηση ήταν η εξής υπάρχουν, ε, τις γνωρίζετε και οι επενδυτές απάντησαν πολύ απλά όχι. 50% δεν είχαν ιδέα τι είναι ένα BIT, διμερής επενδυτική συμφωνία, μόνο 10% είχαν χρησιμοποιήσει στην επαγγελματική τους δραστηριότητα μια τέτοιου είδους συνθήκη. Δυστυχώς η έρευνα δεν ρώτησε κατά πόσο είχε σχέση με την επίλυση διαφορών η επαγγελματική δραστηριότητα ή με την επενδυτική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει μας δίνει μια πρώτη ιδέα ότι θα, είμαστε, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί κατά πόσο είναι σημαντικές οι επενδυτικές συμφωνίες κοινωνία ε, όπως πολλοί υπέρμαχοι αυτών υποστηρίζουν. Δεν είναι βέβαια παράλογο να πει κανεί ότι οι επενδύτες ε, από το 2000 και μετά έχουν γνωρίσει πολύ καλά τις επενδυτικές συμφωνίες γιατί αυξάνει το αριθμό των ε, ε, μηχανισμών επί, των, της, επί, επίλυσης διαφορών ε, και επειδή βέβαια υπάρχουν και κάποιες διατάξεις προεγκατάστασης ή μετά την εγκατάσταση που συμπεριλαμβάνουν κάποιο στοιχείο απελευθέρωσης και μπορεί να είναι πιο σημαντικό για τις επενδυτικές αποφάσεις. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι μια έρευνα που να είναι πιο πρόσφατη. Θέλουμε μια δειγματοληπτική έρευνα μεταξύ επενδυτικών που έχουν ε, υπογράψει επενδυτικές συμφωνίες με πτυχές απελευθέρωσης και για τη σημασία των επενδυτικών αυτών συμφωνιών ε, σε σχέση με το πόσο αποτελεσματικές ήταν αυτές οι συνθήκες. Ένας Αμερικάνος συνάδελφος ε, ζήτησε μία τέτοιου είδους έρευνα μεταξύ 75 πολυεθνικών, πόσο γνώριζαν δηλαδή τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και πόσο σημαντικές ήταν κατά την απόφαση επενδύσεων στο εξωτερικό εκπληκτικά τα αποτελέσματα. τα, κάποιοι τα γνώριζαν πολύ καλά, αλλά ήταν λίγοι αυτοί και οι περισσότεροι δεν γνώριζαν τις επενδυτικές συμφωνίες και γνωρίζαν, δεν, δεν γνώριζαν κατά πόσο έπαιζαν ένα σημαντικό ρόλο κατά στο κατά πόσο θα έκαναν επενδύσεις στο εξωτερικό οι αμερικανικές πολυεθνικές. Υπήρχε αυτοί υπήρχαν αυτές οι περιπτώσεις, ήταν πολύ σπάνιε. Να σκεφτούμε λοιπόν για μια στιγμή ότι η επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα θα δώσει σημαντική πρόσβαση ε, παραπάνω από αυτή που θα δίνει η Κίνα στο εγγύ μέλλον. Νομίζω ότι κατά πόσο θα γίνει αυτό είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων ή όχι, αλλά τέλο πάντων είναι μια πιθανότητα. Ακόμη και αν υπάρχει τέτοιου είδου σενάριο, δεν θα υπάρξει σοβαρό αντίκτυπο στην απόφαση των Ευρωπαίων επενδυτών για το πόσο θα επενδύσουν στη Κίνα ή το αντίστροφο. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να πει ότι υπάρχουν και άλλοι έμεση τρόποι αντίκτυπου των επενδυτικών συμφωνιών στις επενδυτικές ροές Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που αναφέρεται συχνά ως βασικό σύνδεσμος, ε, τεχνικό, είναι τέλος πάντων ε, η διασφάλιση κάποιου πολιτικού κινδύνου. Δεν ξέρουμε όμως κατά πόσο σε αυτό βοηθάει η επενδυτική συνθήκη. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει αποτέλεσμα στις ε, στην επενδυτική συμπεριφορά ο τρόπος με τον οποίο έχει, ο η επενδυτική συνθήκη μια, ένα τέτοιο είδους αποτέλεσμα είναι αυτή η διασφάλιση του πολιτικού ε, ε, κινδύνου. Σε μία λοιπόν ε, έρευνα που έκανα πριν από κάποια χρόνια σε τομέα υψηλού κινδύνου, οι απαντήσεις ήταν ότι ποτέ σχεδόν δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις επενδυτικές συμφωνίες. Υπάρχει βέβαια ε, και ένα γερμανικό ε, παράδειγμα που αποτελεί εξαίρεση, αλλά να σας πω αυτή η σημαντική σημαντικοί εταίροι της αγοράς τι έλεγαν, ε, Βρετανικός φορέας είπε ότι μπορεί η επενδυτική συμφωνία να μας δίνει κάποια καθοδήγηση, αλλά δεν είναι ε, πάρα πολύ σημαντική στην αποφασή μας. Και αυτό απάντησαν και πολλοί άλλοι φορείς. Ε, και η Παγκόσμια Τράπεζα είπε το ίδιο πράγμα. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, οπότε να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πάρα πολύ σπάνια, ακόμη και σε, πολιτικό, σε, σε, σε επίπεδο εκτίμηση του πολιτικού κινδύνου, ε, σπάνια λαμβάνονται υπόψη αυτέ οι επενδυτικέ συμφωνίε. Αυτό σημαίνει ότι παρά το γεγονό μια τέτοια επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα μπορεί να έχει αποτέλεσμα στη νομική δομή των επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. θα είναι πολύ σπάνιο να έχει κάποιο αντίκτυπο ε, στον προορισμό ή στον όγκο των επενδύσεων αυτών αν οι εμπλεκόμενοι φορεί των διαπραγματεύσεων αυτών μεταξύ, μον, μεταξύ αυτών και εσείς ε, έχουν πολύ πολιτικο, πολύ, πολλούς πολιτικούς λόγους για τους ε, οποίους ε, η γραφειοκρατία θα έπρεπε να ξεκινήσει με μια πολύ μακροχρόνια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει χρηματοδότηση και αν το πολιτικό κεφάλαιο μια τέτοια διαδικασίας δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλα σημαντικά θέματα κατεπήγοντα πολιτικές σχέσεις δηλαδή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ε, μεταρρύθμιση ε, του, του, του, της, ε, της επένδυσης πόρων που έχουμε κάνει για τις επενδυτικές αυτές συμφωνίες. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον αρνητικό και είναι πραγματικά αμφίβολη η συνεισφορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Ε, όποτε κάνουμε έρευνε στη δική μου εκλογική περιφέρεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθω δεν ξέρουν ποιο είναι ο Πρωθυπουργό τη Αγγλία, ε, όχι να ξέρουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε με εκπλήσουν μερικά από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι είναι οι διμερεί επενδυτικέ συμφωνίε. Λοιπόν, επόμενος ομιλητής είναι ο καθηγητής ε, Wen Hua Shan. Ήδη τον ε, παρουσίασα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί εγώ πρέπει να φύγω και θα αναλάβει την Προεδρία ο Χέλμουντ. Um, um, Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που με καλέσατε να συζητήσουμε τις ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Κίνας στο πλαίσιο των, ε, της προοπτικής των ομιλιών για μια διμερή επενδυτική συνθήκη. Ε, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα το ότι βρίσκομαι εδώ. Γιατί πριν από λίγα χρόνια είχα δημοσιεύσει στο Journal of World Trade μία ομιλία για τις ε, επενδυτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και είχα προτείνει μία διμερή επενδυτική συνθήκη. Το ότι 12 ε, χρόνια αργότερα βρίσκομαι εδώ λοιπόν είναι για μένα μεγάλη χαρά γιατί βλέπω ότι συζητούνται σοβαρά αυτά τα θέματα. Είμαι ο μόνος νομικός ε, στο πάνελ. Θα περιοριστώ λοιπόν ε, στις νομικές πτυχές του θέματος. Θα προσπαθήσω να καλύψω τρία θέματα. Πρώτον, ποιο είναι το τρέχον νομικό πλαίσιο για τις επενδυτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Δεύτερον, γιατί πρέπει να εξετάσουμε την προοπτική μιας διμερούς επενδυτικής συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και τρίτον, ποια είναι τα βασικά νομικά θέματα στις δυνητικές συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη διμερή επενδυτική συνθήκη. Το πρώτο θέμα λοιπόν, ποιο είναι το τρέχον νομικό πλαίσιο. Η απλή απάντηση είναι ότι υπάρχουν διάφορα κομμάτια από νομοθετικές διατάξεις από διάφορες χώρες. Υπάρχουν στοιχεία διεθνούς δικαίου και στοιχεία εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Υπάρχουν διαμερείς συνθήκες μεταξύ ε, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Κίνας και ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συμφωνία Συνεργασίας Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει η, Επιτροπή, υπάρχει Σύμβαση για την επίλυση διαφορών ICSID, η Σύμβαση MIGA, οι συμφωνίες του ΠΟΕ Η σύμβαση ΜΙΓΑ εξειδικεύεται στο να παρέχει εγγυήσει για τις επενδύσεις και οι συμφωνίες ε, του ΠΟΕ περιλαμβάνουν κάποιες επενδυτικές ρήτρες για το εμπόριο και για τις υπηρεσίες συγκεκριμένα και υπάρχει και η συμφωνία TRIMS που έχει σχέση με το εμπόριο και υπάρχουν κάποια στοιχεία όπως το τοπικό περιεχόμενο, το ισοζύγιο πληρωμών Υπάρχουν ε, και ε, νομοθετικές διατάξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών. Όπως επίσης και η κινέζικη νομοθεσία ε, παίζει ρόλο. Αυτό είναι το τρέχον νομικό πλαίσιο. Όταν μιλάμε για το διμερές νομικό πλαίσιο, οι πιο σημαντικές συνθήκες είναι αυτές μεταξύ Κίνας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι πλήρης όμως. Έχει υπογράψει η Κίνα 26 διμερείς συμφωνίες, δεν καλύπτεται η Ιρλανδία και μόνο 23 είναι λειτουργικές. Δεν καλύπτονται λοιπόν και άλλες τρεις χώρες. Επίσης, δεν υπάρχει συνέπεια μεταξύ των συνθήκων. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η πρόσβαση στη διεθνή διαιτησία. Υπάρχει διαφορετικό επίπεδο προστασίας για αυτές τις ε, διμερείς επενδυτικές συνθήκες. Στις περισσότερες από αυτές τις διμερείς συμφωνίες προσφέρεται πλήρης κάλυψη για τη διεθνή διατησία επίλυση διαφορών. Σε κάποιες ε, μόνο τα θέματα αποζημίωσης μπορούν να επιληθούν από την διεθνή διατησία. Διαφορετικά η πρόσβαση είναι περιορισμένη και σε άλλες διμερείς συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία συνένεση για να προσφύγουν σε διαιτησία. Το επίπεδο λοιπόν προστασίας και το επίπεδο ανοίγματο είναι διαφορετικό σε αυτές τις διμερείς συμφωνίες και αυτό δημιουργεί διακριτική μεταχείριση ανάλογα με την χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία πρόκειται. Επίσης υπάρχει περιορισμένο αποτέλεσμα της ρήτρας του πλέον ευνοουμένου κράτους αυτή η ρήτρα θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισότιμο πεδίο και το επίπεδο προστασίας που θα προσφέρεται σε όλες τις χώρες θα μπορούσε να είναι ισότιμο. Όμως σύμφωνα με τα διάφορα συμβούλια διατησίας, δεν είναι ίσο το επίπεδο εφαρμογής της ρήτρα του πλέον ευνοουμένου κράτους. Κάποιες συμφωνίες συνεργασίας έχουν ευρία κάλυψη, αλλά ε, δεν ε, δημιουργούν ε, νομικές υποχρεώσεις και στις δύο πλευρές, άρα δεν προσφέρουν ασφάλεια στις επενδύσεις και δεν ενθαρρύνουν τις αμοιβέ επενδύσεις. Με μια σύντομη λοιπόν επισκόπηση του τρέχοντος νομικού πλαισίου μπορεί να πει κανείς ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο δεν είναι πλήρες, δεν είναι συνεπές, ιδίως όσον αφορά το διεθνές νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει συνέπεια. Είτε είναι πολύ γενικές οι διατάξεις, είτε πάρα πολύ εξειδικευμένες. Η συμφωνία Ε, μπορεί να είναι πολύ γενική και κάποιες άλλες διατάξεις να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένες. Ε, περνάω στο δεύτερο σημείο που είπα ότι θα αναπτύξω. Γιατί να εξετάσουμε μία διμερή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας μια διμερή επενδυτική συνθήκη. Καταρχήν ενισχύει την διμερή νομική προστασία. Θα μας εξοικονομήσει κόστος, θα καλύπτεται πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καλύπτεται και η Ιρλανδία. θα καλύπτονται και οι τομείς που δεν καλύπτονται τώρα, δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών και θα υπάρξει δυνατότητα απελευθέρωσης της πρόσβασης στην αγορά αν συμπεριληφθεί η πρόσβαση στην αγορά ε, σε αυτή τη διμερή επενδυτική συνθήκη. Η Κίνα παίρνει ιδιαίτερα σοβαρά τις διεθνείς δεσμεύσεις της ε, μετά την ένταξη στον ΠΟΕ. Έχει αλλάξει η Κίνα και δεν ισχύει αυτό το οποίο στο παρελθόν μπορούσε να προσάψει κανείς στην Κίνα. Και μετά την ένταξη στον ΠΟΕ, η Κίνα θα βοηθηθεί να προάγει τις μεταρρυθμίσεις της και αυτό θα έχει επιπτώσει και στις συνθήκες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα βελτιωθούν τα νομικά συστήματα σε εσωτερικό επίπεδο και στην Κίνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει δοκιμαστικά μια τέτοια σημαντική διμερή επενδυτική συνθήκη και θα επωφεληθεί από αυτό και θα βελτιωθούν ε, οι νομοθετικές διατάξεις ε, και στην Κίνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διευκολυνθεί επίσης η διαπραγμάτευση πολυμερών επενδυτικών συμφωνιών, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα διάκυνται θετικά προς κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε για δυνητικέ συνομιλίε ε, για διμερή επενδυτική συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, ποια είναι τα βασικά ζητήματα. Είναι η απελευθέρωση των επενδύσεων, η προστασία των επενδύσεων, η επίλυση διαφορών και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η απελευθέρωση των επενδύσεων είναι το πιο σημαντικό θέμα των δυνητικών συνομιλιών ε, διότι στο παρελθόν η Κίνα ποτέ δεν συμφώνησε σε υποχρεώσεις προ της εγκατάστασης. Πάντοτε είχαμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα με αυστηρές διατάξεις και δεν δεσμευόταν η Κίνα σε μεταχείριση εθνική μεταχείριση πριν από την εγκατάσταση του επενδυτού. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει απελευθέρωση των επενδύσεων. Δυσκολίες υπάρχουν, διότι δεν έχουν ε, εμπειρία καμία από τις δύο πλευρές ε, σε τέτοιες ε, συνομιλίες απελευθέρωσης επενδύσεων. Μπορούμε να έχουμε ένα θετικό κατάλογο και ένα αρνητικό κατάλογο. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο, γιατί έχω ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο ομιλία μου. Ε, όχι, μην διακόψετε, συνεχίστε, αλλά προσπαθήστε να κλείσετε την ομιλία σας. Είναι λοιπόν ε, κάτι που θα απαιτήσει πολύ χρόνο γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους ισχυρούς και αδύναμους τομείς και να δουν ε, πού μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και πού μπορούν να ανοίξουν στον υπόλοιπο κόσμο. Η προστασία των επενδύσεων είπαμε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Η επίλυση διαφορών ε, είναι άλλο ένα θέμα, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εμπειρία σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της υπεράσπισης των υποθέσεων ποιος θα φέρει το οικονομικό βάρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, θέλω να πω εν κατακλείδη, είναι ε, βασική επενδυτική εταίροι με τεράστιο δυναμικό. Και μια διμερής επενδυτική συνθήκη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας θα βοηθήσει να ενισχύσει αυτήν την εταιρική σχέση και να ε, υλοποιηθεί στην πράξη αυτό το δυναμικό το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν στις διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβάνοντας την πρόσβαση στην αγορά και την απελευθέρωση των επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Wen Hua Shan. Πέντε λεπτά μας έχουν μείνει και θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να μας πει πώς θέλει να χειριστεί το θέμα. Γιατί εσείς μας εκφράσατε την κινέζικη θέση. Η ευρωπαϊκή πλευρά όμως ήταν ξεκάθαρη. Δεν χρειαζόμαστε συνθήκη για τις επενδύσεις. Διμερή συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να σας δώσουμε το λόγο για να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση έχει ως εξή. Πριν από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είχαμε τον καταμερισμό των ευθυνών. Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν ε, δεσμεύσει πρόσβαση στην αγορά στι ε, συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου ω τμήμα του ΠΟΕ και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Όμω δεν είχε την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται για επενδυτική προστασία. Η επενδυτική προστασία, λοιπόν, αυτή η πτυχή καλυπτόταν από τα κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την Ιρλανδία καλύπτονται από διμερή εμπορική, ε, επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Το, το θέμα του κατά πόσο είναι χρήσιμο ή όχι να έχουμε μια επενδυτική συνθήκη με έναν τόσο στρατηγικό εταίρο ε, όσο η Κίνα έχει στρατηγικο ε οσο η ληφθεί και η απόφαση είναι θετική όλα τα κράτη-μέλη από την Ιρλανδία που δεν έχει διαπραγματευτεί καμία ε, επενδυτική συμφωνία διμερή αποφάσισαν πριν από πολύ καιρό ότι μπορεί να είναι χρήσιμε οι επενδυτικέ ε, συμφωνίε. Τώρα όμω έχουμε δύο επιλογέ στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Πρώτον, μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα ω έχουν. Έχουμε όλα τα κράτη-μέλη που θέλουν να προστατεύονται, προστατεύονται. Οι συμφωνίε δεν είναι όλε οι ίδιες, υπάρχουν πολλέ διαφορέ. Ή εκμεταλλευόμαστε το γεγονό ότι μπορούμε να δράσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα, σε διαδοχικές συνόδους με την Κίνα, είναι ότι έχει νόημα να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την αρμοδιότητα αυτή για να διαπραγματευτούμε μια επενδυτική συνθήκη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι απλώς μια παγίωση των ε, υπαρχουσών διμερών ε, συμφωνιών, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι πολλά από τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα το, σήμερα το απόγευμα διάρκειες από πλευρά επενδύσεων, μειονεκτήματα σε σχέση με την κινέζικη αγορά, δεν θα μπορούσαμε να τα καλύψουμε. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι αν θέλουμε όντω να φτάσουμε μέχρι την πλήρη διαπραγμάτευση μια συμφωνία με την Κίνα, πρέπει να συμπεριλάβουμε στοιχεία πρόσβαση στην αγορά. Γιατί πιστεύουμε ότι αν συμπεριλάβουμε τα στοιχεία αυτά, θα έχουμε ένα πολύ πιο ισχυρό εργαλείο που θα μειώσει το κόστος για τους οικονομικούς εταίρους και θα δώσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ολοκλήρωσης ε, της, ε, ε, των οικονομιών Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και της Κίνα. Βέβαια έχουμε κάποια εκρεμή ζητήματα σε σχέση με τις λεπτομέρειες και την ουσία. Από την κινέζικη ηγεσία στη Σύνοδο είχαμε θετικά μηνύματα, συμφώνησαν με τη διατύπωση ότι διαπραγμάτευση επενδυτική συμφωνίας πρέπει να καλύψουν όλα τα σημεία που αποτελούν ανησυχία και για τι δύο πλευρέ. Ε, με βέβαια ένα άνοιγμα διαπραγμάτευσης για την πρόσβαση στην αγορά. Θα θέλαμε λίγο περισσότερο, λίγο σαφέστερες ενδείξεις από την πλευρά της ε, κινέζικης κυβέρνησης όσον αφορά την προθυμία τους να συζητήσουν αυτό το θέμα της πρόσβασης στην αγορά. Και όταν λάβουμε αυτές τις ε, σαφέστερες ενδείξεις, βέβαια και εμείς θα παρουσιάσουμε την, τις, διαπραγματευτικές οδηγίες για ε, τη συνθήκη αυτή. Είπαμε προηγουμένως ότι χρειάζεται και μία αξιολόγηση αντικτύπου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία επιλογή, τα στοιχεία της ε, πρόσβασης στην κινέζικη αγορά να συνεισφέρουν όντως στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καλύπτουν κάποια από τα μειονεκτήματα που έχουμε εμείς εντοπίσει στην επενδυτική μας σχέση με την Κίνα. Θα σταματήσω γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα έρθετε το θέμα από δικής μου πλευράς. Πότε θα είναι διαθέσιμη η αξιολόγηση αντικτύπου και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το λέω, αλλά και επειδή μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας, για το κοινό θα θέλαμε να ξέρουμε πότε θα έχουμε αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου και από τη δική μου προσωπική εμπειρία θα ήθελα να πω ότι οι επενδύσεις μερικές φορές μπορεί να παρακολύουν την οικονομική ανάπτυξη σε μερικούς τομείς ε, γιατί μειώνουν την ανταγωνιστικότητα κάποιων κλάδων. Και από την Γερμανία αυτή είναι η εμπειρία μου. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν προς ποια κατεύθυνση και με ποια κριτήρια ε, μπορούμε να προβούμε σε αυτή την επενδυτική συμφωνία και γι' αυτό το λόγο θα ήμουν υπέρ επενδυτική συνθήκης παρά το γεγονός ότι η Οξφόρδη μας είπε σήμερα ότι είναι αμφισβητήσιμο κατά πόσο έχει νόημα να έχουμε μια τέτοιου είδους ε, συμφωνία. Ίσως μπορείτε να μας απαντήσετε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης αντικτύπου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ε, είπα, το έχουμε δρομολογήσει, είμαστε σε επαφή με τι κινεζικέ αρχέ για να καταλάβουμε καλύτερα τι προθέσει ε, και των δύο πλευρών. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την ε, σύστασή της για τις διαπραγματευτικές οδηγίες, θα υπάρξει και κοινοποίηση της αξιολόγησης αντικτύπου Για την ώρα όμως επισήμως δεν υπάρχει αξιολόγητη αντικτύπου γιατί δεν έχει εγκριθεί από το σώμα των επιτρόπων ακόμη. Όσον αφορά τώρα το σχόλιο σας για τις επενδύσεις. Προφανώς όταν λέμε ότι η επένδυση είναι κάτι το θετικό, πάντοτε έχουμε υπόψη μας ένα συνολικό θετικό αποτέλεσμα, ένα συνολικό θετικό αντίκτυπο όπως και σε όλες τις ε, διαδικασίες ε, απελευθέρωσης υπάρχουν τομείς ε, που κερδίζουν περισσότερο από άλλους και τομείς οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο. Προφανώς αυτή είναι η έννοια, αυτό είναι το νόημα της πρόσβασης στην αγορά. Θέλουμε να καλύψουμε τους πιο ευαίσθητους τομείς τους οποίους θα μεταχειριστούμε με περισσότερη προσοχή ως προς την πρόσβαση στην αγορά. Για το ερώτημα τώρα που θέσατε για την εφαρμογή των νόμων και των κανόνων, η διμερής επενδυτική συμφωνία ή κανόνες επενδύσεων ε, δεν επιτρέπουν παρέκκληση από την ε, εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Ένας επενδυτής που έρχεται να επενδύσει στην Ευρώπη πρέπει να ε, σέβεται την ε, νομοθεσία στα κράτη-μέλη και βέβαια αυτήν την αρχή θέλουμε να τη διατηρήσουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Δυστυχώς ε, είμαστε στην κατάσταση την οποία φοβόμουν όταν οργανώσαμε την ακρόαση. Δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία που οργάνωσε την ακρόαση αυτή, παρά το γεγονός ότι και το δεύτερο μας πάνελ ήταν πάρα πολύ ε, καλό και έθεσε διάφορες προκλήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, δύο ε, ομιλητές που ήταν εδώ και θα ήθελα να ολοκληρώσω την ακρόαση, να σας ευχαριστήσω για τη χρήσιμη συμμετοχή σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απάντησε στις ερωτήσεις μας. Συμπεραίνω ότι ήταν ε, μια πολύ επικοδομητική και αποτελεσματική ε, συζήτηση, ένας διάλογος ε, με αξία για μας. Είμαι πεπισμένος ότι στις περαιτέρω εργασίες μας αλλά και στην εποπτική ομάδα των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να ε, ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει αυτή τη επενδυτική συνθήκη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Κίνας και θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη υπομονή και ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σα, για τη συμμετοχή σας, να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, γιατί ξεπεράσατε και το ωράριό σα. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όλες οι παρουσιάσεις σε μερικές ημέρες ε, στον ε, ιστότοπο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι διαθέσιμες και θα έχετε όλη τη δυνατότητα να ε, διαβάσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις παρουσιάσεις των καθηγητών. Επίσης μου ζητούν να ενημερώσω τα μέλη και το προσωπικό της Επιτροπής μας ότι η επόμενη συνεδρίαση ε, θα λάβει χώρα στις 26 Νοεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα και στις 27 Νοεμβρίου ε, και 9 ε, με 12.30 και 3 με 6.30 και θα έχουμε και ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.